Buongiorno a tutti, prendete posto che cominciamo perché siamo già un po' in ritardo. Ξεκινούμε με λίγη καθυστέρηση, λέει η Πρόεδρος. Και θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της Μεσής Διατάξεως, η οποία, όπως πάντα, σας έχει ήδη μοιραστεί. Και αν έχετε κάποια παρατήρηση ή ένσταση, να την υποβάλλετε, ιδάλλως θεωρείτε ότι εγκρίνεται η μερσία διάταξη. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις της Προέδρου, εγώ θα ήθελα κυρίως να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας την 3η 27 Μαρτίου. Θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή των Μεταφορών για τον μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης. Δυνάμει του άρθρου 51. Και γι' αυτό και ήθελα να σας το επενθυμίσω. Και αυτό επίσης να ληφθεί υπόψη για το χρονοδιάγραμμα που θα έχουμε. Πάμε τώρα ή στο τέταρτο σημείο τη ημερησίας διατάξεως που είναι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. θα το συζητήσουμε και με χαρά μας παρευρίσκεται στην αίθουσα κύριος Ντανιέλ καλέ που ασχολείται με τις ε, ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά θα εκπροσωπεί στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Για το ευθύ αμέσω θα δώσουμε την σκητάλη στον ε, εισηγητή για να μας ε, παρουσιάσει τις προτάσεις του ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο αναφέρεται ως κόσμο για την περίοδο 2014 και 2020 περιλαμβάνει τα, τις πτυχές ε, του προγράμματος που λύγει το 2013 και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του προηγούμενου προγράμματος όπως, όπως η ενέργεια, η οικοκαινοτομία και ούτω καθεξής συνεχίζονται στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Παραμένουν λοιπόν τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας του 7ου προγράμματος πλαισίου. Αυτό αφορά για παράδειγμα τα διοικητικό άχθο, τα χρήματα οικονομικά μέσα για το ίδιο κεφάλαιο και για την ε, χρηματοδότηση και το ε, Ευρωπαϊκό Δικτύο Επιχειρήσεων. Καλώς ορίζουμε ιδιαίτερα ότι το, πρόγραμμα, ε, το παλιό πρόγραμμα συνεχίζεται στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, 20, όπως και προγραμματιζόταν. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε στην Ένωση την ανταγωνιστικότητα. Οι Ευρωβουλευτές θα συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Το... Ο προπολογισμό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί ε, μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε 1,25 ε, δισεκατομμύρια. Αυτή η αύξηση ήταν πραγματικά κάτι το απολύτως απαραίτητος γιατί από τις θετικέ μας εμπειρίες με τον προηγούμενο πρόγραμμα SIP ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και την κρίση που διανύουμε. Θα ήθελα να υποβάλω και κάποια, ε, κάποιες προτάσεις βελτίωσης. Το πρόγραμμα COSME θα πρέπει να εστιαστεί σε θέματα ανταγωνιστικότητας. Οι πολιτικοί στόχοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και μερικές προσαρμογές. Τέσσερις στόχοι υπάρχουν. Δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, το, το ότι τονίζουμε το θέμα της ε, βιωσιμότητας αποτυπώνεται και στους μεμονωμένους στόχους. Είναι σημαντική η πολιτική προτεραιότητα, αλλά δεν θα έπρεπε να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πρότασης, γιατί έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ το πρόγραμμα αυτό, δεδομένου και του περιορισμένου προϋπολογισμού, να επικεντρωθεί σε ένα βασικό στόχο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αλλά αυτό θα ισχύει για όλους τους τομείς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. και έτσι πέρα από την υποστήριξη της βιωσιμότητας ε, θα πρέπει όλα αυτά να υποστηριχθούν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Εκεί, για παράδειγμα, έχουμε 6 δισεκατομμύρια για την καθαρή ενέργεια. 7,2 δισεκατομμύρια για τις καθαρές μεταφορές. Ε, και ούτω καθεξής. Ο όρος ε, βιωσιμότητα μπορεί όμως και μόνο σε θέματα ε, κλιματικής ε, βιωσιμότητας οι στόχοι ξεπερνούν κατά 3,5 δισεκατομμύρια τον προϋπολογισμό του κόσμου. Αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τι σημαίνει αυτό. Θέλουμε ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά με βιώσιμο τρόπο στο πρόγραμμα. Και όταν κοιτούμε την ε, βιωσιμότητα υπό το οπτικό αυτό πρίσμα, τότε δημιουργείται μια σωστή συνάφεια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους οικονομικούς τομείς θα πρέπει να λαμβάνουν ίσες ευκαιρίες. Και δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο, το δεδομένο ότι συμπεριλαμβάνεται πλέον και τουρισμό στο πρόγραμμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Im Rahmen des Einzel... Also, wir wissen, dass Tourismus... Äh, Ξέρουμε ότι ο τουρισμός ε, έχει υπογραμμιστεί ιδιαίτερα στο ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας και η σημασία του στην Επιτροπή ΙΜΚΟ υπέβαλα και μία έκθεση για το πώς μπορούμε ε, στην Ευρώπη να διαμορφώσουμε τον τουρισμό, γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται και πέρα από τα εθνικά σύνορα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το προσέξουμε. Σίγουρα υπάρχουν έργα στον τομέα αυτό, που, όπου μπορούμε να συνδράμουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα του τουρισμού, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να πληρούνται και οι σχετικές προϋποθέσεις ασφαλώς. στον τομέα του τουρισμού ε, έχουμε 131 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών σχεδίων έχουμε μόνο 87 εκατομμύρια. Αυτό που είναι σημαντικό και αυτό θα πρέπει να αποτελεί το βασικό μας μήνυμα είναι ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν το καταφέρουμε αυτό, τότε θα δημιουργήσουμε και νέε θέσει εργασία, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Στα πλαίσια των σχετικών πρωτοβουλειών θα πρέπει να τονιστεί και να υποστηριχθεί η μεταφορά των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την εξαγορά ε, επιχειρήσεων από πιο δυναμικές επιχειρήσεις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι σε μη αποτελεσματικέ μεταφορές επιχειρήσεων θα χαθούν ε, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή πώς θα καταφέρουμε να υπάρξει μια συνέχεια στις επιχειρήσεις, όταν για παράδειγμα οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχουν την ευκαιρία ε, να συνεχιστούν μέσω άλλων μελών της οικογένειας. Θα πρέπει να είναι σαφής η διάκριση μεταξύ του προγράμματος κόσμου και ορίζοντας 2020. Για παράδειγμα, στο πρώτο πρόγραμμα COSME μιλάμε ε, για την, τα προϊόντα και για την παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ε, παραγωγικότητας των πόρων. Όλες αυτές οι πτυχές αποτελούν, θεωρώ, απόρρια της καινοτομία, η οποία δεν βασίζεται απαραίτητα στην έρευνα, αλλά ίσως και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών. Άρα θα πρέπει να δούμε την ε, καινοτομία και κατά πόσον ίσως δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME, γιατί λείπουν πόροι. Θα πρέπει με τον απλούστερο τρόπο ε, να διευκολύνουμε την ε, εισαγωγή και την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα αυτό. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ υψηλές οι απαιτήσει που τίθενται για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάτσουμε από κοινού με τους συναδέλφους για το πρόγραμμα Ορίζοντας, Ορίζοντας 2020 για να δούμε πώς θα μπορούμε να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν την πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πόρους του προγράμματος COSME θα πρέπει να το κάνουμε αυτό και θα πρέπει να δούμε μήπως θα πρέπει καλύτερα να αφήσουμε το πρόγραμμα ορίζοντας 2020 για αυτό που προορίζεται για την κοινοτομία. Οι δείκτες ε, ε, με τους οποίους μετράται η επιτυχία του προγράμματος θα πρέπει επίσης να τύχουν επεξεργασίας γιατί σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ποσοτικούς και όχι τόσο ποιοτικούς ε, δείκτες προκειμένου να μετράμε αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για, για το διοικητικό άχθος. Δεν έχει νόημα ίσως τόσο πολύ να κοιτάμε πόσες ε, προϋποθέσεις έχουν καταργηθεί. Ίσως θα έπρεπε να δούμε καλύτερα κατά πόσο έχει μειωθεί το κόστος ε, συμμετοχής για μια μικρομεσαία επιχείρηση και να ορίσουμε μια ποσοστία μείωση για παράδειγμα. Και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί μια σωστή ε, σκέψη. Το ανώτατο όριο που ορίζεται θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό σε ό,τι αφορά τις, ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. οι πιστώσει για τις μη καινοτομικές ε, ε, επιχειρήσεις πάνω από τα 50.000 ευρώ ουσιαστικά δεν καλύπτονται από κανένα από τα δύο προγράμματα παρά το γεγονός ε, ότι υπάρχουν ε, ανάγκες οι οποίες ε, ξεπερνούν τις προσδοκίες σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ θα μπορούσαν να σημειωθούν βελτιώσεις. Και έτσι θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε και μεγαλύτερες ε, επενδύσεις τις οποίες χρειαζόμαστε. Κατά έβδομο, η, τα χρηματοπιστωτικά ε, μέσα θα πρέπει να καλύπτουν αδυναμίες των εθνικών συστημάτων. Και σε ό,τι αφορά διασυνοριακές ε, πιστώσεις. Η ζήτηση περιορίζεται υπερβολικά σε εθνικά όρια και χρειαζόμαστε ναι, ναι, κλείνω, Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσεις σε τοπικές αγορές. Η ευρωπαϊκή αγορά, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα ήταν ακριβώς αυτό στο επενδυτικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Τα είπα κάπως περιεκτικά αλλά νομίζω κάτι τέτοιο περιμένετε πάντα από τον εισηγητή, να δίνει κάποιες καινούργιες σκέψεις και ευχαρίστω να ακούσω και αυτά που έχουν να πούν και οι συνάδελφοι αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή, κ. Καλέγια Κρέσπο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά να σήμερα να σα απευθύνω το λόγο και να σα ε, παρουσιάσω ε, το πρόγραμμα Κόσμο προ την Επιτροπή σα, διότι από την 1η ε, Φεβρουαρίου έχω αναλάβει αυτό τον τομέα ω Γενικό Διευθυντή, αλλά ήδη, ήδη επί ένα έτος ε, ασχολούμαι με τι ΜΜΕ ω ειδικό απεσταλμένο και θα συνεχίσω αυτό να το κάνω. Επομένω, γι' αυτό σα λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταδειχθεί το πόση σημασία αποδίδουμε στην πολιτική για τι ΜΜΕ. Έχω εδώ κάποιες διαφάνειες με τις οποίες μπορώ να σας παρουσιάσω τους στόχους και τα βασικά σημεία γραμματός κόσμου. Στο πρώτο, στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε πόσο σημαντικές είναι οι ΜΜΕ για την ευρωπαϊκή οικονομία και αυτό θα πρέπει να είναι η αφετηρία οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονομία, μια που έχουμε 23 εκατομμύρια ΜΜΕ, ε, που είναι 99% δηλαδή των ευρωπαϊκών εταιριών. Και πρόκειται για την ε, μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας θέσεων εργασία. Δύο από τις, ε, σε κάθε τρει θέσει εργασία είναι από τι ΜΜΕ. Για κοιτάξτε τα στατιστικά. 85% όλων των νέων θέσεων εργασία <clears throat> ε, έχουν δημιουργηθεί από τι Ευρωπαϊκέ Επιτροπέ. Οπότε γι' αυτό λέμε που για τι τη ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει επομένω να υπάρχει μια πάρα πολύ δυναμική πολιτική για να τι υποστηρίξει. Δεύτερη διαφάνεια. Είναι όμως και δυνατός κρίκο, διότι η οικονομική κρίση έτσι ε, έχει χτυπήσει πάρα πολύ ε, ποιες επιχειρήσεις αυτές. Ήδη είπαμε ότι έχουμε 23 εκατομμύρια 24 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι, 10% του εργατικού δυναμικού. Επομένως πρόκειται για ένα μέσο έλλειμμα του ΑΕΠ 7% και μιλάμε για 80% του ΑΕΠ ε, για το επίπεδο των, του, του, του, του χρέους. Και επίσης έχουμε τα παγκοσμία προβλήματα τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στις ΜΜΕ, άρα βλέπετε πώς ε, τις έχει χτυπήσει αυτή. Ποια είναι τα προβλήματα τα οποία τώρα αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, πρώτα-πρώτα ε, δεν έχουν ρευστότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο σήμερα ε, έχουν. Έχουν αυτό το, την έλλειψη ρευστότητα. Credit crunch, το είναι τρίτον δηλαδή, αυτών των ΜΜΕ, που ζήτησαν δάνειο από τράπεζα τελικά δεν πήραν τη χρηματοδότηση που θέλανε. Ή του απάντησαν αρνητικά, τους είπαν δεν μπορούμε να σα δώσουμε αυτά όσα ζητήσατε. Και είναι μεταξύ 500.000 και 700.000 και πρόκειται για αυτά τα νούμερα ε, επιχείρησεων που το πρόβλημα αυτό. Δεύτερον, προσβασιμότητα στι νέε αγορέ. Μόνο μία στι τέσσερι των ευρωπαϊκών ε, ΜΜΕ κάνει απευθείας εξαγωγές στις άλλες ε, ε, αγορές στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο μία στις 8, 13% εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει κρατικό πρόβλημα για να εξαγάγουν. Τελευταίο, αλλά σημαντικό τώρα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας εξηγήσω. Πρόκειται για την γραφειοκρατία. Το πόσο δύσκολο είναι μία ΜΜΕ να συμμορφωθεί με όλα όσα συνεχώς επιτάσσονται από την νομοθεσία, διαδικασίες, δηλώσεις, διατυπώσεις. Μεγάλο το πρόβλημα. Και εγώ, όποτε έχω με παιχνίδες ΜΜΕ, μου λένε, κάνε κάτι, δεν πάει άλλο. Με όλα αυτά που μας ζητάνε. Τα γραφειοκρατικά επομένως. Εμείς τι κάνουμε για αυτό το πρόβλημα. Κάνουμε το κόσμο, το πρόγραμμα κόσμο και αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε είναι η ΜΜΕ να ενταχθούν και να καλυφθούν από τις δημοσιογραφικές προοπτικέ. Και οπότε, το διορθωτικά ταμεία, τα χρηματοδοτικά μέσα, όλα αυτά να έχουν και μία πτυχή, μη, μη, έψιλον αλλά κατά δεύτερο λόγο επίσης αυτό το οποίο προτείνουμε είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα επί τούτου για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη που να καλύπτει τις μία έψιλον. Πρόκειται για το κόσμο. Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη για τις οικονομικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για 2,5 δις ευρώ προϊκοδότηση και όπως ακριβώς ο κύριος Κρόιτσμαν έχουμε το παρουσιαστικό αποτέλεσμα επειδή σε σχέση με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τα προγράμματα SIP. Έχουμε αυτά τα τέσσερα προγράμματα λοιπόν των ΜΜΕ και θα πρέπει να δούμε πώ θα σα βοηθήσουμε να έχουν προσβασιμότητα στη χρηματοδότηση, πώ θα μπορούσαν να προσβασιμότητα ή στι αγορέ, να δούμε κατά τρίτο λόγο πώ θα βοηθηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και και επίση να δούμε τι θα γίνει, πώ θα έχουν καλύτερε συνθήκε να κάνουν τη δουλειά του. Θα καλύψουμε αυτά τα τέσσερα προγράμματα. Πρώτα-πρώτα, χρηματοδότηση. 1,4 δι είναι η χρηματοδότηση Δύο βασικά χρηματοδοτικά μέσα, ε, χαμηλέ εγγυήσει με μία προκοδότηση 1,4 ε, ευρώ και εμεί του προτείνουμε περισσότερε εγγυήσει για δανειοδότηση. Γιατί αυτό, διότι στα μεγαλύτερα κράτη-μέλη, όταν πηγαίνουν στι τραπέζε για να προσφύγουν για υποστήριξη <clears throat> και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αυτό του χρειάζεται. Οπότε, σήμερα τα δικά μα στατιστικά υπάρχει το αποτέλεσμα της μόχλευσης. Για κάθε ευρώ έχουμε 30 επιπλέον ευρώ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία για τα επιπλέον. Επίση, τώρα όσον αφορά τα venture capital funds, το κεφάλαιο του οικονομικού κινδύνου, διότι τώρα στο SIP έχουμε 2,2 δις ευρώ, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί με 200, 350 συγγνώμη, εκατομμύρια των επενδύσεων. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι, το, αποτέλεσμα, το, το, η επίδραση τη μόχλευση είναι πάρα πολύ σημαντική. 1,4 δι επομένω όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα. Και κατά δεύτερο λόγο, το δεύτερο τμήμα, δεύτερη προτεραιότητα του πράγματο είναι πώ θα υπάρχει καλύτερη απόδοση στι αγορέ. Και γι' αυτό θέλουμε να επιδρώσουμε την προσοχή μα στο πώ θα παρέχονται υπηρεσίε προ αυτέ τι επιχειρήσει για να μπορούν αυτέ να επεκτείνουν δραστηριότητά του. Και όταν εξάγουν, μπορεί να έχει θέσει εργασίε καινούριε, μπορεί να κάνει και δομέ. Όμω έχουν ένα σωρό προβλήματα και αυτό χρειάζονται την βοήθεια χρειάζονται κατάρτιση, εκπαίδευση, ενημέρωση, πληροφόρηση και επομένω για να έχουν καινούριου πελάτε και εταίρου θα πρέπει να του δώσουμε τι ευκαιρίε. Έχουμε το επιχειρηματικό ευρωπαϊκό δίκτυο και που του δίνει αυτέ τι υπηρεσίε. Και γι' αυτό και επίση θα θέλαμε να έχουμε αναβαθμισμένη υποστήριξή του. Με αυτό το δίκτυο επιχειρήσεων της Ευρώπης αυτό είναι καλό θεμέλιο και έχουμε και επίσης αυτή το πρόγραμμα μικρές εταιρείε, σαν μεγάλο κόσμο 600 τέτοια κέντρα πληροφόρηση έχουμε, συνδέονται με τα επιμελητήρια, με τους φορείς των ε, επιχειρήσεων και έχουμε και 3.000, 3.000 προσωπικό για να βοηθάει. Επίσης, θα συνεχίσουν, θα συνεχίσουμε με κάποια στοχευμένη βοήθεια και ας πούμε να, έχουμε αυτή την υπηρεσία, αυτό το γραφείο στην Κίνα για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να λύσουν τα προβλήματά τους σε κάποιες οικονομίες. Το Κοινοβούλιο έριξε την ιδέα. Πρόκειται για μια πιλωτική δράση. Και πρέπει να σας ευχαριστήσω. Γιατί χάρη σε αυτό το γραφείο λαμβάνουν πάρα πολύ σημαντική βοήθεια οι επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικό. Άρα χρειάζεται δίκτυο να κάνουμε χαρτογράφηση. Δεν θέλουμε τώρα να κάνουμε επικάλυψη στις δουλειές, αλλά χρειάζεται υποστήριξη προς τις μηνύσεις των τρίτων. Το πώ θα βοηθεί η επιχειρηματικότητα κάτι το οποίο είναι ένα πρόβλημα σημαντικό στην Ευρώπη. Άνοιξτε μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία, όλο ένα και λιγότεροι Ευρωπαίοι θέλουν να λάβουν κινδύνους. Όταν και λιγότεροι θέλουν να ξεκινήσουν τη δική του επιχείρηση. Και αν κάτσετε και συγκρίνετε με ΙΠΑ και Ασία, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη όσον αφορά τη συγκρότηση, την ίδρυση εταιριών και επιχειρήσεων. Οι νέοι, εδώ είναι το σημαντικό στοιχείο, χάρη στο Κοινοβούλιο, ξεκίνησε αυτό το έρασμος για τους νέους επιχειρηματίες που και έτσι μπορούν να περάσουν έξι μήνες σε κάποιον πιο έμπειρο επιχειρηματία και θα πρέπει αυτή η πρωτοβουλία να ενισχυθεί. Πρόκειται για πρόγραμμα που έχει σημειώσει επιτυχία. Αλλά θα βλέπουμε και τι γίνεται και με τι γυναίκε επιχειρηματίε. Έχουμε λοιπόν, το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκτυο. Η πρέσβυρε τη επιχείρηση είναι ένα άλλο παράδειγμα, που δραστηριοποιούμαστε σχετικά με αυτό σε 22 χώρε και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Προκειμένω για άλλο ένα τομέα ή στον οποίο μπορεί να βοηθήσει το κόσμο. Τέταρτη προτεραιότητα, το πώς θα βελτιωθεί το πλαίσιο το επιχειρηματικό το κλίμα το επιχειρηματικό για να δούμε τι θα κάνουμε απλούστευση μείωση γραφειοκρατίας πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει στην εφαρμογή της, του νομοθετήματος για τις μικρές ε, επιχειρήσεις θα ε, βελτιωθεί θα διευκολυνθεί η υλοποίηση των αποφάσεων Ας πούμε, η μεταφορά των επιχειρήσεων δεν διευκολυνθεί. Μια δεύτερη ευκαιρία που μπορεί να δοθεί στις επιχειρήσεις και με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να έχουμε ανταλλαγή εμπειριών για τις ε, άριστες πρακτικές και εδώ πρέπει να θυμηθούμε τους απεσταλμένους ΜΜΕ. Κάθε χώρα έχει έναν και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούμε την πρόοδο αυτής της πρωτοβουλίας. Το κόσμο επομένως μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εργαλείο. Εργαλείο για να βοηθήσει στην υλοποίηση αυτών των μέτρων. Και στην εισήγηση του κ. Κρότσμαν ανέφερε διάφορα, μεταξύ των οποίων είπε για το πρόβλημα στον τουρισμό, για την ειδική νομική βάση. Μας είπαν οι νομικοί ότι για το ΣΥΠ χρειάζεται ειδική νομική βάση. Για να καλύψουμε όμως τα πάντα. Δεύτερον, για τη μεταφορά των επιχειρήσεων. Σημαντικό αυτό που θα χρηματοδοτηθεί και επίση μα ανέφερε τη σχέση με την υπόθεση ορίζουν 2020 και αύριο έχουμε ένα εργαστήριο πάνω σε αυτό. Οπότε και θα περιμένουμε να μας βοηθήσει να ξεκαθαριστεί η σχέση των δύο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα μας είπε για την ομάδα Στόιμπερ ο κύριος ε, Κρόιτσμαν ναι και για τους δείκτες επομένως για τα κριτήρια θα βοηθήσει αυτή η ομάδα επίσης είπε ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα του επίπεδου δανεισμού το μία και τώρα κατακλείδη θα πρέπει να σας πω με την τελευταία μου διαφάνεια το μήνυμα το μήνυμα είναι η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ότι η αποτελεί υψηλή προτεραιότητα η πολιτική τη ΜΜΕ και θα πρέπει τώρα περισσότερο ποτέ να κινητοποιήσουμε πόρου να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε οι που είναι τα θύματα της δημοσιογραφικής κρίσης να μπορέσουν να βγουν από την κρίση σαν πρωταγωνιστές, πρωταγωνιστές του ξεπεράσματος της κρίσης. Επομένως, ας βοηθήσουμε τις ΜΜΕ και αυτό το κάνουμε χέρι-χέρι με το Κοινοβούλιο εκτός όπως έχουμε υποσχεθεί. Grazie. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο πρώτος παρόν εδώ τουλάχιστον ο ο Thank you so much. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι συμφωνούμε ότι μία από τι βασικές προκλήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μα είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις αγορές και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Οι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά ελκυστικέ. και νομίζω ότι ο Γενικός Διευθυντή ε, μας έκανε μια πολύ εμπεριστατωμένη εισαγωγή για το ζήτημα αυτό. Μ' αρέσει η γενική ιδέα να γίνει ένα streamline των κοινοτικών προγραμμάτων και θέλουμε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 να προβλέψουμε καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά την πρόταση COSME, μου αρέσει πολύ αυτή η εξορρόπηση που έγινε μεταξύ των, των μεγαλεπίβολων διορατικών προτάσεων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος ε, με και το συνδυασμό με βραχυπρόθεσμους στόχους όπως είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαιο και σε δανεισμό. Είναι όμως χαλεπές οι οικονομικές συνθήκες, γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι μόνο 0,2% του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και των συζητήσεων για τον προπολογισμό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τον προπολογισμό του κόσμου. Προσβλέπω σε ε, εμβριθή συζήτηση με τον κύριο Κρόισμαν και τους υπόλοιπους και οδησηγητές. Πιστεύω ότι σε αρκετές περιπτώσεις μπορούμε να βελτιώσουμε την έκθεση. Για τον τουρισμό, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει να επιταψιλεύσουμε τόσα κονδύλια. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Τι γίνεται. Ε, νομίζω ότι άλλοι τομεί είναι πολύ σημαντικοί γιατί θα πρέπει να ενισχύσουμε ένα τομέα ει βάρος άλλων. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η σωστή μέθοδο να μεροληπτήσουμε υπέρ ενό τομέα. Και αν είναι να ενισχύσουμε ένα τομέα, υπάρχουν άλλοι με πολύ καλύτερε προοπτικέ ανάπτυξη από ότι ο τουρισμό. Τι γίνεται με την εξαγωγή υπηρεσιών. Η εσωτερική αγορά υπηρεσιών είναι μια καινούργια αγορά και υπάρχουν εκεί πολύ τεχνητοί φραγμοί για τις εξαγωγές επιχειρήσεων, σε ε, υπηρεσιών, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές πρωτοβουλίες που θα εξυπηρετούν όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε μια κατάσταση όμως όπου οι τράπεζες είναι προσεκτικές και εξαιρετικά επιφυλακτικές και απρόθυμες να δανείσουν θα πρέπει εμείς να δούμε πώς θα βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κεφάλαιο για να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Άκουσα ότι μόνο το 1 τρίτο, το, το 1 τρίτο συγγνώμη, των επιχειρήσεων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το δανεισμό που χρειάζονται. Μ' αρέσει πάντως ε, η εξορρόψη που έγινε μεταξύ του Long Guarantee Facility και του Equity Facility στο κόσμο. Πιστεύω πάντως ότι ο προπολογισμό του COSME είναι σχετικά χαμηλός σε σχέση με την επιρροή που θα έχει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τον απότερο σκοπό μας, δηλαδή μεγαλύτερη μόχλευση των κοινωτικών κονδυλίων και να πιάνουν τα χρήματα τόπο εκεί που δίνονται. Θα πρέπει τα χρήματα να είναι πολύ κοντά στι επιχειρήσει, ε, κοντά στην επιτόπια διαχείριση. Επίση, ε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και του διοικητικού άχθους. Χρειαζόμαστε πραγματικούς αυτούς στόχους μείωσης της γραφειοκρατίας. Καθημερινά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με την ε, θέσπιση νέων οδηγιών συμβάλλουμε στην ενίσχυση της γραφειοκρατίας. Γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για μείωση τη γραφειοκρατία σε ένα τομέα. Χρειαζόμαστε σαφεί, καθαρού στόχου μείωση τη γραφειοκρατία. Ό,τι αφορά την πρόσβαση στι αγορέ, θα πρέπει να προβλέψουμε συμπληρωματικέ δομέ και προγράμματα. Αυτό είναι κεφαλόδου σημασία για να βοηθήσουμε τι τις ε, ευρωπαϊκέ μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, να διεκδικήσουν νέα μερίδια αγορά. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και αργότερα. Και τέλος, δεν θεωρώ ότι το πρόγραμμα COSME που έχει τόσο ε, μικρό προϋπολογισμό θα πρέπει να διευρυθεί και σε άλλες χώρες, στις υποψήφιες δηλαδή χώρες. Να βοηθήσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις των υποψήφιων χωρών, αλλά ε, όταν χώρες, ε, κάποιες χώρες δεν θέλουν να ε, ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να αξιοποιούν τα κοινοτικά κονδύλια που στόχο έχουν την ενίσχυση της κοινοτικής ανταγωνιστικότητας. Μην ξεχνάτε ότι ε, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τα, τα χρήματα των φορολογουμένων των χωρών μελών. Ας προσέξουμε λοιπόν ποιες χώρες θα ωφελήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Έχουν ε, συμπεριληφθεί πολύ στο κατάλογο μιλητών. Θα ήθελα να κλείσω τώρα το κατάλογο και να θερμοπαρακαλέσω τους αγορητές να περιοριστούν στο τρίλεπτο. Ο κύριος Ρουμπίχη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που ο κύριος Κρόιτσμαν ε, ε, τόνισε τα απαραίτητα στοιχεία της έκθεσης αυτής, γιατί το θέμα είναι πολύ απλά πώς ε, θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Η κρίση του χρέους μας αναγκάζει να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με, ε, και προϋποθέσεις πλαίσιο στα οικονομικά Το θέμα είναι πώς ε, θα μπορέσει να γίνει η επανακεφαλοποίηση των ε, κρατών μελών, όχι μόνο των τραπεζών και αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί το ποσοστό ιδίου κεφαλαίου στον ε, κλάδο αυτό είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις ΗΠΑ και δεν υπάρχει φυσικά χωρίς περαγκαιότητα πίστοση για κάποια επιχειρήση και μετά από τις προσπάθειες ε, επενδύσεις φαίνεται ότι δεν προκύπτουν οι ανάλογοι υψηλοί μισθοί. Όπως είπε και ο υπουργό ε, Οικονομικών της ε, Μίκλος, θα πρέπει να αφήσουμε τα χρήματα εκεί όπου είναι πλέον παραγωγικά και αυτό ισχύει για τις πιο νέες επιχειρήσεις. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με τις ιδέες και ξέρουμε ότι οι νέοι επιχειρηματίες έχουν πολύ μεγάλη απόδοση για κατά μέσο όρο 49 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δίκαιος ο μισθός για τους επιχειρηματίες αυτούς. Και γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο το σύστημα των προμηθειών να ξαναδιαμορφωθεί. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι όταν ξεκινάει μία νέα επιχείρηση, το κόστος αυτό που καταβάλλεται στην αρχή να επιστρέφεται μόνο εν μέρη. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει καλύτερη τέτοια απόσβεση. Στην Αμερική ε, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόστους ε, των εξόδων μπορεί να δηλωθεί και να αποσβεθεί ως κόστος. Ε, στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι έτσι και η φορολογία είναι μεγαλύτερη. Οδηγεί λοιπόν σε πιστώσεις στις επιχειρήσεις για να διακόψουμε λοιπόν αυτό το φαύλο κύκλο θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως ε, για τις νέες ε, επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να προβλέψουμε κάποιες φορολογικές ε, απαλλαγές και να κοιτάξουμε πιο πολύ τις μισθούς που καταβάλλονται. Γιατί ποιος, ποιος έχει απόδοση για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει όταν ξεκινάει μια καινούργια επιχείρηση από ένα νεαρό επιχειρηματία, συμμετέχει στον ρίσκο, αν θέλετε, πέρα τον επιχειρηματία και η οικογένειά του και οι φίλοι του σε πολλές περιπτώσεις, ενώ οι τράπεζες μένουν άτεγκτες. Και αν τελικά συμβεί κάτι, αυτοί είναι που ζημιώνονται και όχι οι τράπεζες. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πριμ για τον κίνδυνο λοιπόν αυτών που διαθέτουν τα χρήματα αυτά και επενδύουν σε μια επιχείρηση. Είμαι εισηγητή ε, για την Επιτροπή Προπολογισμού για την έκθεση COSME. Οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όμως σε πολυεθνικό επίπεδο θα πρέπει να λάβουν την υποστήριξή μας ε, γιατί αυτές είναι που τελικά χάνουν από την παγκοσμιοποίηση και νομίζω ότι το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση θα έπρεπε να εξετάσει το πώς θα μπορούσε να υποστηρίξει στις δραστηριότητε τους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τις κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβιάσεων. Κοιτάξαμε και την περίπτωση της Microsoft και πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλες αυτές, ε, όλες αυτές οι κυρώσεις, όλα αυτά τα πρόστιμα θα πρέπει να διατίθονται στο πρόγραμμα COSME. Και φυσικά οι ταμείοι χρησιμοποιηθέντα κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη θα μπορούσαν επίσης να προστίθενται στο πρόγραμμα αυτό. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Τεχνολογία. Σκοπός του είναι η διάδοση της γνώσης. Προκειμένου να είμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο ανταγωνιστικοί. Αυτά περιλαμβάνονται και στην ατζέντα της Λισαβόνας και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το πρόγραμμα COSME για να καλυφθούν και το ποσοστό, το υψηλό ποσοστό ανεργίας που έχουμε στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρούμπιχ. Πολύ σημαντική η παρέμβασή σας και για τις αναφορές που κάνατε στον προϋπολογισμό. Αλλά αν όλοι μακρηγορούν τόσο πολύ, δεν πρόκειται να ολοκληρώσουμε σήμερα την ημερήσια μας διάταξη. Κύριε Μέρκης, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, και τον ε, Γενικό Διευθυντή για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και την πολύ εμπεριστατωμένη επισκόπηση που μας έκανε. Θα θέλαμε κάπως πιο διεξοδικές όμως ε, εξηγήσεις για το, το σύνδεσμο του κόσμου με το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα ορίζοντας 2020 γιατί αν καταφέρουμε να καινοτομήσουμε με καλύτερο τρόπο θα είναι πιο εύκολη και η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Πρώτα χρειαζόμαστε ένα προϊόν που πουλάει και ένα καινοτόμο προϊόν πουλάει πολύ καλύτερα από ένα γενικό προϊόν. Συνήθως έχουμε είτε ένα καινοτόμο προϊόν είτε ένα πολύ παραδοσιακό προϊόν όπως για παράδειγμα μια και Έχουμε εδώ την πρόεδρο από την Ιταλία, τα πολύ ωραία ε, ιταλικά design που κάνουν το γύρο του κόσμου και είναι και ευπόλυτα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτή η σύνδεση μεταξύ των δύο. Σε ό,τι αφορά την καινοτομία που παράγει επιχειρήσεις ε, και που αναβαθμίζει τις επιχειρήσεις, τι κάνει το κόσμο για τις επιχειρήσεις αυτές. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους ε, που λένε ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα μεσούς της χρηματοπιστωτικής κρίσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα με τους κανόνες, γιατί έχουμε πολλούς και διάφορους κανόνες. Έχουμε πληθώρα κανόνων και διατάξεων που ουσιαστικά εμποδίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και εμποδίζουν και την πρόσβασή τους ε, στις ε, άλλες αγορές πλην των εθνικών, των εγχώριων αγορών. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι προτιμούμε να δημιουργούμε νέες ευκαιρίε παρά να καταργούμε εμπόδια και φραγμούς που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν φραγμοί στην δική μας την αγορά. Δεν υπάρχει εσωτερική ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της πιστοποίησης είναι προβληματικό για πολλέ επιχειρήσει, ιδιαίτερα για φαρμακευτικά προϊόντα. Πώς θα πάρουν πιστοποίηση σε άλλες αγορές. Οι προδιαγραφές ασφάλειας. Όλες οι προδιαγραφές ε, μερικές φορές δημιουργούν ανυπέρβλητους φραγμούς. Κάντε μας λοιπόν μια επισκόπηση της συνολικής προσέγγισης ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και όχι μόνο τη προσέγγιση του κόσμου, γιατί με ενδιαφέρει μια πληρέστερη εικόνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μέρκη. Το λόγο κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και του συναδελφού Κρόιτσμαν, αλλά και από το Γενικό Διευθυντή. Έχω τρει σύντομε παρατηρήσει τι οποίε θα ήθελα να αναφέρω, αλλά θα ήθελα να τονίσω εκ νέου αυτά που είπε και ο συνάδελφο Ρουμπίχ. Ότι το Α και το Ω είναι το κεφάλαιο κινδύνου για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Νομίζω ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να παρέχουμε τις ε, ανάλογες ε, διευκολύνσεις. Ε, συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει να δουν κίνητρα και στα κρατημέλη για φορολογικές απαλλαγές σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, αν και δεν μπορεί να διαμορφωθεί από ευρωπαϊκό συνάδελφοι, εμείς πάντα ελπίζουμε να δημιουργήσουμε τις σωστές ε, προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα ε, λόγια δεν ακολουθούνται από πράξεις. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που πλήττονται πιο πολύ. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα, ότι καταβάλουν προσπάθειες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έχουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από συστάσει της Επιτροπής Στόιμπερ, αλλά μέχρι ότου εφαρμοστούν αυτά, μέχρι ότου υπάρξουν αποτελέσματα, παίρνει χρόνια. Για παράδειγμα, η απλοποίηση στα κράτη-μέλη, δεν ξέρω πόσο καιρό το συζητάμε το θέμα αυτό. Για τα λογιστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν ισχύουν τα ίδια που ισχύουν για τους μεγάλους ομίλους. Θέλαμε λοιπόν ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από ό,τι ξέρω τα πράγματα έχουν κολλήσει στο Συμβούλιο. Δεν μπορώ παρά να απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει πίεση προκειμένου να κινηθούν τα πράγματα. Ιδάλλως δεν πρόκειται να μας εμπιστευτούν πλέον καθόλου όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι και άλλα πολλά μπορώ να αναφέρω τους τοχογράφους και ούτε καθεξής. Για την ενίσχυση τώρα κατά δεύτερον των επιχειρήσεων. Ασφαλώς και συμφωνούμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες είναι τεράστιο δυναμικό των επιχειρηματιών, των γυναικών. Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να δραστηριοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά πολιτικές προτεραιότητες, προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία. Όταν προσπαθεί κάποιος ε, στην Ευρώπη να δημιουργήσει μια επιχείρηση και αποτυχάνει, θεωρείται αποτυχημένος. Ενώ στις είπα δεν υπάρχει η ανάλογη νοοτροπία. Νομίζω ότι μέσα από τα προγράμματά μας μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και κατά τρίτον, τελευταίο θέμα σε ό,τι αφορά την απλοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται μελέτες αντικτύπου. Γίνονται εδώ και πολλά χρόνια εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά μπορούμε να επικρίνουμε, αλλά αυτό που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί την εξή πολιτική πλέον. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει ανάλογα με τον ορισμό στην Ευρώπη, εξαιρούνται από τις ε, προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός και αν αποδεχτεί ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Άρα αυτή η αλλαγή σε ό,τι αφορά την εξαίρεση ή μη, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, θετική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος, και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Χέρτσοκ. Κυρία Χέρτσοκ, Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι σύντομη, αλλά όμω έχω δύο θέματα δικά μου και άλλα δύο για την κυρία Παντιζετό, που είναι ισχυρό και δεν μπορεί να παρασταθεί. Δεν, δεν θέλω να πω κάτι για το κόσμο, αλλά θα πρέπει να σας συγχαρώ για την ψυχική εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ σημαντική πρόκληση η ψηφιοποίηση για τις ΜΜΕ και πάλι συγχαρητήρια και με χαρά μας να βοηθήσουμε στην επίση προγράμματος. Τώρα κάτι δεύτερο που θέλω να σας πω για δικό μου ότι ό,τι κάνετε σε επίπεδο νησιακό θα πρέπει, θα πρέπει λέγω να έχει τη, βάση του στη δράση των 100 μερών. Επομένω, θα πρέπει και εμεί να θέλουμε έκκληση στα να μην τα παρατήσουν όσον αφορά την πολιτική διαμήνυση στην Ουγγαρία. 83% του προγράμματο έχει υλοποιηθεί. Και να δούμε τι θα γίνει με τον κόσμο. Ξέρετε τι πρέσβευε για τον κόσμο. Να σας πω ότι είπε και δυσκιώδη δηλαδή συγκεντρία. Λέει εκείνη ότι το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και ο τελικός στόχος είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητε που υπάρχουν για ανάπτυξη γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την Ευρώπη ΜΜΕ και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το, το, το η κρίση ρευστότητα γιατί οι τράπεζε αρνούνται τι πιστώσει, αρνούνται τα δάνεια υποφέρουν επομένω από την έλλειψη κεφαλαίου μήψεων. Αυτό επομένω είναι πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να εκκρεμεί και άρα θα πρέπει να έχουν ευκολότερη προσβασιμότητα ή στην χρηματοδότηση και αυτό είναι σημαντικό να του ξαναδώσουμε καινούργια όθηση και σε αυτέ και στην απασχόληση. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποια συνοδευτικά διαρθρωτικά μέτρα. Να έχουμε αυτά τα δίκτυα, το οποίο είναι κάτι το αναγκαίο, ούτω ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί παγκόσμια. και θα πρέπει να υπάρχει μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προγραμματιστούμε μακρόπνοα. Αυτά τα προβλήματα απασχολούν όλες τις ΜΜΕ και χρειάζεται η κατάρτιση των επιχειρηματιών για να ενταχθούν στα δίκτυα. Να τους δώσουμε τα όπλα για να μπορέσουν να σταθούν στην παγκόσμια οικονομία, το κόσμο επισημαίνει το πού χρειάζεται ευρωπαϊκή, ενωσιακή παρέμβαση, αλλά δεν λέει το πώ θα γίνει αυτή η παρέμβαση, Ιδίω όσον αφορά την διεθνοποίηση, την πλαισίωση των δράσεων που θα χρειαστούν για να βγουν στην παγκόσμια αγορά επιχειρήσεις και γίνεται τώρα και άλλοι λέει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και το θέμα της ισότητας ευκαιρία των φίλων και τονίζει ότι για να γίνουν πιο διεθνείς όπως είπε η ΜΜΕ θα πρέπει και να κάνουμε για την γραφειοκρατία. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία πρεσβεύει η κυρία ω ως σκιώδης εισηγήτρια. Grazie, Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κύριο Οντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις προτάσεις που κατέθεσε. Σε ό,τι αφορά τους γενικούς στόχους, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει κανένα αποχρόν λόγο να συμπεριλάβουμε και τον τουρισμό. Αναφέρατε τη νομική βάση, αλλά νομίζω ότι είναι περί τη συμπερίληψη του τουρισμού. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση, άκουσα τι παρατηρήσει για τα προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την απλοποίηση των κανόνων λογιστικής. Αναφέρθηκε ένα σχόλιο του κ. Σόιμπλε και όταν είπε ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα λογιστικά. Νομίζω ότι είναι ανόητο αυτό. Ε, θα πρέπει απλώς να ενημερώνονται σωστά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνει κάποια απλούστευση. Ε, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση. Το πρόβλημα της ε, περιπλοκότητας δεν οφείλεται στη λογιστική, αλλά στην υπερβολική ρύθμιση, στις διατάξεις φορολογικές, κοινωνικές. Είμαι από τις χώρες που είναι πρωταθλήτριες των ρυθμίσεων και των κανονισμών που δεν εφαρμόζονται οι χώρε θα πρέπει να πλουστεύσουν την νομοθεσία του. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που ένα επίτροπος θεσπίζει μια διάταξη, υποβάλλει μια οδηγία, τον υποχρεώνουμε να, καταργήσει, ναι, τον υποχρεώνουμε να καταργεί δύο. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η πρόταση για να ξεκινήσουμε με τη μείωση τη γραφειοκρατίας από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με την, με την ηλικία των στελεχών, των ε, υψηλόβαθμων στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι περισσότερες είναι πολύ μικρές και δεν ενδιαφέρουν. Ε, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη ε, έμφαση και στα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια για να σπυρώσουν καλύτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, σε ό,τι αφορά τι πολύ μικρέ επιχειρήσει. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το ποσοστό θνησιμότητα αυτών των πολύ μικρών νέων επιχειρήσεων. Γιατί πολλέ ε, μικρέ επιχειρήσει εξαιτία έλλειψη ιδιοπόρων ε, χαμηλή πρόσβαση στο δανεισμό και επειδή ε, αφήνονται στο έλεος τους τα πρώτα χρόνια, πεθαίνουν στα σπάργανά τους πολλές μικρές επιχειρήσεις. Και εδώ θα πρέπει να διαδραματίσουν καλύτερο ρόλο τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια. Επίσης, χρειαζόμαστε έναν σωστό κοινωνικό διάλογο μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Γιατί το, το, η συνθήκη τη Λισαβόνα μα επιτρέπει να έχουμε πανευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο για να διασφαλίσουμε ένα πρόσφορο κοινωνικό κλίμα και στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Οντί, Το λόγο του κύριος Λάγκεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την παρουσίαση που μας έκανε ο Γενικός Διευθυντής σχημάτισε την εντύπωση ότι τώρα μόλι ξεκινάμε μια πολιτική για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είμαι χρόνια ολόκληρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θυμάμαι ότι ο Επίτροπο Μπάγκεμαν, που εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1999, ήδη τότε είχε ένα σχέδιο, τότε που μιλούσαμε για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και χρόνια από το 1990 φαίνεται ότι δεν έχει κάνει καμία πρόοδο σε αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ο αριθμό. Ε, ε, όλες οι προτάσεις ε, έγιναν, απορρίφθηκαν. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι γίνεται με τον ορισμό. Διατίθεται, προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πρόγραμμα αυτό να συμπεριλάβει και τις μικρόμεσες επιχειρήσεις. Ο συνάδελφος Μπέντς μίλησε για τους φορολογούμενους. Ε, από ό,τι θυμάμαι, εδώ και 15 χρόνια τα μέσα των Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων δεν αυξάνονται. Καταρχάς επειδή υπάρχει πολύ υψηλή γραφειοκρατία και κατά δεύτερον επειδή οι μικρομεσαίες ε, τράπεζες προτιμούν να συνεχίζουν μόνες τους και είναι τόσο ελάχιστη η διαφορά των επιτοκίων. Και κατά τρίτον επειδή οι ετούντες ε, δεν έχουν ε, δυνατότητα να καταλάβουν τι γίνεται τρίτη ερώτηση στο θέμα του κεφαλαίου κινδύνου. Εδώ μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά πράγματα. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σχετικές προτάσεις, θα πρέπει αυτό να γίνει βάση των εμπειριών των τελευταίων δύο δεκαετιών. Εγώ πιστεύω αναφέρθηκαν πολλές ε, μεμονωμένες ε, διατάξεις από την κυρία Νίμπλερ, την κυρία Ρούμπιχ, τον κύριο Μπέντσεν. Αναρωτιέμαι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το σωστό σημείο αφετηρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με σοβαρότητα. Με όλη την νοσταλγία που τρέφουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. βλέπω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λείπει το απαραίτητο, ο απαραίτητος μύτος, αν θέλετε, που θα μας οδηγήσει. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Ευαγγελία Πράγμα. Και τώρα, τον λόγο έχει ο κύριο Σοντή, ο οποίο προηγουμένω μίλησε λιγότερο χρόνο από όσο δικαιούται προηγουμένω. Αλλά ξανέχετε το λόγο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, το, το, ξέχασα, ξέρετε να ξεχάσω το θέμα της προσημότητας στις ε, αγορές ε, του κρατικού τομέα. Έχουμε, ξέρετε, ένα ψήφισμα με ισχυρή πλειοψηφία του Γιώργου Μακρύδη ε, ή προ τον κύριο Μακρύδη τέλο πάντων, ο οποίο είχαμε πει ότι θα πρέπει στον ΠΟΕ να ζητήσει παρέκκληση για την προσβασιμότητα στι κρατικέ αγορέ. Και ακατανόητο το, το, γιατί ήρθε σε εκείνη τη στάση. Το τι γίνεται όσον αφορά την ποσόστοση, το ποσοστό που δικαιούνται από τις δημόσιες συμβάσεις, ε, τις δημόσιες αγορές, τις κρατικές αγορές. Ε, οι, οι μη μη εψιλών. Έχετε το λόγο. Κυρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κρότσμαν και τον κύριο Γενικό Διευθυντή που έρθει να μας μιλήσει. Μας τα είπε τόσο διεξοδικά. Ξέρετε, ήμουν επιχειρηματία. Πολύ καιρό. Και εμεί θέλω να σα πω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι θα πρέπει να βιαστούμε, να κατεβάσουμε ταχύτητα, διότι έχουν πάρα πολλέ επιχειρήσει, οι οποίες ματώνουν, ματώνουν, φιλορωούν όσον αφορά το ότι δεν ξέρουν από τη μια μέρα στην άλλη τι θα απογίνουν. Πρέπει να ενεργήσουμε ταχύτητα. διότι δεν ξέρουν τι, τι, τι θα τις βρει, τι τις περιμένει. Από μια μέρα στην άλλη. Επίσης θα πρέπει κάτι να κάνουμε και για τους νέους. Όντως, οι νέοι για πολύ καιρό όντως δεν ανελάμβαναν πρωτοβουλίες. Και δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν επομένως και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τόσο ώστε να αρχίσουν να ρισκάρουν. Να μπορούσαν να έχουν μια επιχειρηματική διαδρομή και σταδιοδρομία επιτυχή. Να δούμε πώς θα γίνει και με τις ε, μεγάλες αγορές όπως Κίνα και Ινδία. Προσοχή γιατί και εκεί τα πράγματα, το κλίμα είναι αρνητικό. Υπάρχουν θέματα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα και επίσης υπάρχουν θέματα με το τι θα γίνει με την κατάθεση των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνία στην Ευρώπη και πολλέ φορέ πρέπει να θα περιμένει πάρα πολύ. έχουμε πάνω σε αυτά τα 2,5 δι ω προοικοδότηση, κάτι το οποίο όμω είναι φραγκοδίφραγκα, διότι είπαμε ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον τη Ευρώπη. Γιατί η συμφωνητική στήλη είναι φραγκοδίφραγκα, εάν κάτσουμε και συγκρίνουμε με αντίστοιχη προοικοδότηση, αντίστοιχα ταμεία τα οποία διατίθενται. Διότι χωρί κεφάλαιο, χωρί πόρου, χωρί προβλασιμότητα στην χρηματοδότηση, αυτό το πρόβλημα δηλαδή, που σήμερα έχουν ε, επιχειρήσεις ε, δεν μπορούν να, να, να, να εμπορευθούν ούτε εντός και κυρίως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Έχει το λόγο επόμενος. Κύριος Κέλλη. Περισσότεροι συνάδελφοι με κάλυψαν. Πάντως ήθελα και εγώ να καλύψω κάποια άλλα θέματα και με τις δικές μου απόψεις. Για τη χρηματοδότηση για το τι ισχύει στη δική μου χώρα. 91% των ΜΜΕ λένε ότι τώρα οι τράπεζες τους δανείζουν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι πριν. 50% των περιπτώσεων λένε όχι. Να, τι ισχύει ή στην Ιρλανδία λόγω της κρίσης. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο δύσκολο είναι να προοδεύσουν οι επιχειρήσεις μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο. Οι προσμετρήσεις στις αγορές επίσης είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. όλο ένα και περισσότερα φυσικά πρόσωπα αρχίζουν να αγοράζουν με το Ιντερνετ. Πάρα πολλέ εταιρείε πάντω δεν μπαίνουν στο Ιντερνετ, άλλε δεν πουλάνε εκτό τη χώρα του. Μεγάλο πρόβλημα. Το Σαββατοκύριακο σε κάποια κυρία η οποία αγόρασε μέσω του Ιντερνετ νηφικό, όχι συγγνώμη, ένα, ένα φόρεμα για τον γάμο της κόρης της. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, ε, αυτό, ακόμα και αν δεν ξαναμπεί στο Ιντερνετ αυτή η κυρία, σημαίνει ότι κάτι έρχεται να αλλάζει. Τώρα, όσον αφορά το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σου πω πάλι τι γίνεται στη χώρα μου. θεωρήθηκε ότι πρόκειται για διασπάθηση των χρημάτων μας. Γιατί αντί για όλα αυτά, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι τα ταμεία να βοηθάνε αυτούς που μείναν χωρίς δουλειά, να τους βοηθάει να στείλουν τη δική τους επιχείρηση. Κατάρτιση, να τους βοηθούν και να μην του υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν δίνονται ποτέ. Πεταμένα λεφτά είναι. Για να το κοιτάξουμε καλύτερα. Επίση, δούμε τι θα γίνει με του νέου επιχειρηματίε και τι γυναίκε. Τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, να μην τα επαναλάβω. Υπάρχουν δυνατότητε που κρύβονται εκεί. Επίση, να δούμε τι θα γίνει με τη γραφειοκρατία. Να τη συγκρατήσουμε, να τη μειώσουμε. Γιατί σήμερα με τα στοιχεία που έχουμε δεν γίνεται τίποτα να κάνουμε κάτι και να αποδείξουμε ότι κάνουμε κάτι για να βελτιωθεί το κλίμα. Ο κύριος Λάγκε επίσης μας ανέφερε κάτι για τις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Νομίζω ότι εδώ έχει νόημα του να έχουμε χωριστή κατηγορία για τις μικρές και, και άλλη κατηγορία και άλλο καθεστώς για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μην προσπαθούμε να τις βάλουμε όλες στο ίδιο καλάθι. Γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μεσαίων. Αυτό είναι σημαντικό από οργανωτική πλευρά. Επίση, τελευταίο, όπω είπε ο κ. Μπένσον, δεν έχει νόημα να τελειθούν χρήματα των φορολογουμένων να βοηθούμε επιχειρήσεις εκτός Ένωση. Να βοηθούμε σε επιχειρήσει που είναι εδώ. Να γίνουν και πάλι ανταγωνιστικέ, να έχουμε πλήρη απασχόληση να είμαστε και πάλι πιο ανταγωνιστικοί και μετά, μετά, μετά να σταματήσουμε και το περιβόλι μας και να βοηθάμε τους ξένους. Πρόεδρος. Φόρντ. Κυρία Φόρντ. Εν συντομία, η μείωση της γραφειοκρατίας θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό μας στόχο. Θα πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ μικρών, μικροσκοπικών αν θέλετε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ίσως να εξαιρεθούν αυτές οι μικροσκοπικές εταιρείε από μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας γιατί πολύ ανησυχώ ότι η νέα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει ελεγχθεί με βάση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν όλη η νέα νομοθεσία να περάσει από ένα τέτοιο έλεγχο αλλά θα πρέπει να κάνουμε και ε, μια αναθεώρηση στο παρελθόν και να δούμε τι μέρος της νομοθεσίας θα πρέπει να θεωρήσουμε σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις πιστώσεις. Ε, ε, συνάδελφοι από πολλές χώρες έχουν καταθέσει σχετικές τροπολογίες για την απελευθέρωση των τραπεζικών κεφαλαίων για τον δανεισμό των επιχειρήσεων. Το υποστηρίζω αυτό, αλλά στο προηγούμενο πρόγραμμα βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες λειτουργήσε το προηγούμενο πρόγραμμα SIP, αλλά σε κάποιες όλες παρουσίασε υπερβολική γραφειοκρατία. Και υπάρχουν άλλα προγράμματα τα οποία λειτουργούν καλύτερα. Άρα θα πρότεινα, εξετάζοντας την δημιουργία νέων εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μήπως θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο απλά εργαλεία σε κράτη-μέλη. Και για παράδειγμα, πρόσφατα πολλές ε, τράπεζες ε, αποταμίευσης μου είπαν ότι θεωρούν τα προγράμματα αυτά υπερβολικά γραφειοκρατικά. Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, για παράδειγμα, σε όλες τις γλώσσες. Υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία για το κεφάλαιο κινδύνου. Αυτό αυξάνεται. Αλλά αυτό προορίζεται ιδιαίτερα για τις ε, μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και τη χρηματοδότηση μεταξύ ομοτήμων. Θα πρέπει και στους τομείς αυτούς να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Ανυπομονώ λοιπόν και προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους και με τον κύριο Κρότμαν και για την έκθεση του κυρίου Ρούμπιχ. Σας ευχαριστώ και η τελευταία παρέμβαση από την κυρία Δελκαστήγιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έφτασα κάπως καθυστερημένα, αλλά είμαι εξοικειωμένη με τις προτάσεις. Έχω διαβάσει τις γραπτές προτάσεις του εισηγητού. Νομίζω ότι είναι τρεις επιτυχίες ε, της πρότασης αυτή. Ε, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι σημαντική, δημιουργεί πρόοδο. Όπως είπε ο κ. Λάγκερ, το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι και παραδοσιακό και ιστορικό. Μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η τελευταία πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι πολύ προοδευτική και από άποψη απλοποίηση, ε, της γραφειοκρατίας, χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Τρία όμω είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να απορροφούν την δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αν επικεντρωθεί σε αυτά τα τρία στοιχεία, θα συμβάλλει πραγματικά στην υπέρβαση των προβλημάτων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι τρεις οι βασικοί άξονες, τρεις οι βασικοί πυλώνες η χρηματοδότηση, δηλαδή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, διοικητική απλούστευση, μείωση τη γραφειοκρατίας και το τρίτο σημείο είναι η εναρμόνιση. Αυτοί είναι οι τρει βασικοί πυλώνε, οι τρει βασικοί άξονε, στου οποίου θα πρέπει να εστιάζεται η κοινοτική δράση. Για τη χρηματοδότηση θα έχουμε ευκαιρία και με τι τροπολογίε μα να εκλεπτύνουμε κάποιε προτάσει τη έκθεση. Πάντω, όπω είπε η κυρία Χόπ, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και να προβλέψουμε για αυτές τη διαφορετική μεταχείριση. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση τη γραφειοκρατίας, τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Αυτό είναι το κατεξοχήν σημείο, η πιο ίσως χρήσιμη πρόταση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 γιατί εξαιτία της ε, διωγγωμένης γραφειοκρατίας ε, πνίγονται στα σπάργανα πολλές ε, και πολύ μικρές επιχειρήσεις και προσπάθειες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν τα φόντα, έχουν το δυναμικό να μετατραπούν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ένας αρτοπιός όταν δημιουργεί το πρώτο το αρτοπείο, στόχο έχει να δημιουργήσει μια λυσίδα αρτοπείων και να προχωρήσει με την καλή αυτή ε, πρόταση για τη μείωση της γραφειοκρατίας θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτυχθούν και να μετατραπούν σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το θέμα της εναρμόνισης, ο τρίτος άξονας. Θέλουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ ε, και την ψηφιακή αγορά έχουμε μια τεράστια δυνατότητα, ε, μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για τις ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Η νομοθετική εναρμόνιση λοιπόν είναι πολύ σημαντική για τα θέματα αυτά. Δεν θα επιμείνω είναι, είναι αυτονόητο ότι το ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο είναι χρήσιμο και θα πρέπει να αναπτυχθεί. Είναι ζωτική σημασία για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο για μια σύντομη απάντηση στον εισηγητή μας, τον κύριο Κρόιτσμαν. Και θα τον παρακαλέσω για κανένα τεταρτάκι να αναλάβει την Προεδρία. Α, γιατί δεν βλέπω άλλον αντιπρόεδρο και για ένα 15 λεπτό θα πρέπει να σας αφήσω παρακαλώ. Ελάτε να αναλάβετε και την Προεδρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτά που μας ανέφερε ο συνάδελφος Λάγκε για το κατά πόσο χρειαζόμαστε καν τέτοια προγράμματα, αυτό αποτελεί ε, και το τελικό ερώτημα του κόσμου. Ε, μήπως ε, θα πρέπει να υπάρχουν εθνικά προγράμματα και τι γίνεται σε, σε διασυνοριακό επίπεδο. Γιατί νομίζω ότι ο μικρός φούρναρης της γωνίας δεν θα ωφεληθεί από το κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό τα πολύ καινοτομικά στοιχεία να περιληφθούν στο πρόγραμμα Ορίζοντες 2020. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε όταν μιλάμε για μείωση της γραφειοκρατίας να συζητάμε και το πώς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους τομείς. Να δημιουργήσουμε σαφείς ορισμούς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί στη μετέπειτα διαδικασία και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ε, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν συνέχεια και του προγράμματος ΣΥΠ. Αυτό είναι σαφές. Δεν μιλάμε για κάτι εντελώς καινούριο. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα συνέχεια ενό παλαιότερου προγράμματο Διαπιστώνω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει έχουν υπερβολικά μικρό ποσοστό ιδίου κεφαλαίου, είπατε κυρία Ρούμπιχ. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν θέματα πρόσβασης της αγορά, πρόσβασης της πιστώσης, κατά πόσον υπάρχει στήριξη, θα πρέπει να υπάρχει στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα εθνικά προγράμματα δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε ασφαλώς, ούτε αυτό είναι ο σκοπός μας. Και γι' αυτό λοιπόν αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να είναι διασυνοριακός χαρακτήρας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και απόδοση των προγραμμάτων αυτών. Ε, εδώ θα περιοριστώ περιέλαβα και τις προτάσεις σας. Θα γίνει και μια κρόαση, θα γίνει και ένα σχετικό σεμινάριο και όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν θα τα συζητήσουμε εις βάθος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρότσμαν. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση για τις εξαιρετικές τους ε, παρατηρήσεις που άγγιξα πραγματικά τα βασικά σημεία, τους κεντρικούς άξονες της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί ως προς τον νευραλγικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ως προς τη σπουδαιότητά τους για την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχει ένα θέμα, ένα ζήτημα με τον ορισμό. Αν θα συμπεριλάβουμε τις μικρές, τις πολύ μικρές, θα γίνει διάκριση μεταξύ μικρών και μεσαίων. Μερικές χώρες είναι να διευρύνουμε το, τον ορισμό, να, να ξεπεράσουμε τους 250 εργαζόμενους, να περάσουμε στους 500 εργαζόμενους. Θα ξεκινήσουμε, θα καταρτήσουμε μια μελέτη, θα κάνουμε μια επισκόπηση κατάστασης και αν κριθεί απαραίτητη μια αναθεώρηση του ορισμού θα το κάνουμε. Αλλά θα πρέπει γι' αυτό να υπάρξει ομοφωνία. Προς το παρόν όμως ε, χρησιμοποιούμε τον ισχύοντα ορισμό. Όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Κρόιτσμαν, το κόσμο δεν είναι το μοναδικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε αντίστοιχα προγράμματα ε, και στο Περιφερειακό Ταμείο. Έχουμε εκεί κονδύλια. Έχουμε στο Ευρωπαϊκό, στο Κοινωνικό, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχουμε στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 κονδύλια για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το κόσμο όμω είναι ένα ειδικό πρόγραμμα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι η συνέχεια του ΣΥΠ και προσπαθούμε να επικεντρωθούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, να επικεντρωθούμε στην προστιθέμενη αξία. Τι προστιθέμενη αξία μπορούμε να επιφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι οι προλαλήσαντες συμφώνησαν ότι μπορούμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο δανεισμό, στη χρηματοδότηση. Μπορούμε να συμβάλλουμε με την απλούστευση, εκεί θα έχουμε θεμενή αξία και άλλο ένα τομέα, άλλος ένας τομέας που μπορούμε να έχουμε προστιθέμενη αξία είναι η πρόσβαση στην αγορά και γενικώ στο πλαίσιο πρόσβαση στο δανεισμό και στη χρηματοδότηση. Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Ήδη χρησιμοποιούμε ε, κάποιες εγγυήσεις δανειακές, διαχείριση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Έχουμε πολύ περισσότερα αιτήματα, πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από, από προσφορά. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals. Έχετε δίκιο κύριε Ρουμπίχ. Θέλουμε περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, γιατί σήμερα έχουμε λιγότερα από, από τα κεφάλαια που είχαμε πριν από μία δεκαετία. Πολύ σημαντικό θέμα, γι' αυτό προτείνουμε να συνεχίσουμε τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα venture capital. Απλούστευση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ένθερμο υπέρμαχο από μένα για την απλούστευση των κανόνων. Όλε οι μελέτε επιπτώσεων θα πρέπει να γίνονται πριν τη θέσπιση νέων προτάσεων. Το τεστ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι απαραίτητο. Και σε μερικές περιπτώσεις να εξαιρέσουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε προβλήματα όμως στο θέμα αυτό, αλλά σίγουρα θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και πριν υποβάλουμε νέους κανόνες, να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν αυτοί οι νέοι κανόνες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νίμπλερ, και την κυρία Φόρτ για τα σχόλιά τους, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το στοιχείο της απλώστευσης στις προτάσεις μας. Πρόσβαση στις αγορές. Είπα, ρώτησαν μερικοί, θα καλύπτουμε μόνο την ενιαία αγορά ή και άλλες τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες, καλύπτονται 17% του ΑΕΠ δίνεται σε κρατικέ προμήθειε και μόνο ένα τρίτο πηγαίνει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μια ποσόστοση. Εμεί δεν έχουμε αντίστοιχη ποσόστοση στην Ευρώπη. Και εγώ λοιπόν διαρωτήθηκα όπως και εσείς, γιατί δεν έχουμε εμείς ποσόστοση. Κατά πάσα πιθανότητα γιατί ε, υπάρχουν περιορισμοί στον Παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου, αλλά ισχύει εξαίρεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά όμως και χωρίς ποσόστοση οι επιδόσεις μας είναι καλύτερες από αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως εξετάζουμε το θέμα και θέλουμε να υποβάλουμε μια πρόταση για πρόσβαση σε δημόσιες προμήθειες τρίτων χωρών και επίση, ε, μια μεταρρύθμιση οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες για να γίνει πιο φιλική αυτή προς τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την ε, συμπερίληψη και των τρίτων χωρών, έλαβα υπόψη τις ε, παρεμβάσεις των κ. Μπένσον και Κέλλη. Θα αγνοήσουμε τελείω το θέμα τρίτε χώρε. Προσοχή, οι, οι, χώρες BRICS για παράδειγμα, ε, το 17% του έπτους θα δώσουν μέχρι το 2030. Δεν λέμε να δώσουμε κονδύλια στις χώρες αυτές, αλλά να διευκολύνουμε τις εξαγωγές προϊόντων των δικών μας χωρών προς τις χώρες αυτές. Γιατί στη Βραζιλία, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Ρωσία έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά ανάπτυξης. Έχουμε το help desk των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κίνα. Ενδιαφέρονται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις ευκαιρίες που θα έχουν στις χώρες αυτές. Πάντω θα συνεχιστεί η συζήτηση και έλαβα υπόψη τα επιχειρήματά σα. Τώρα, ποια είναι η διάκριση μεταξύ του προγράμματο Ορίζοντα 2020 και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ορίζοντα 2020 ε, στηρίζεται στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, όχι μόνο όμω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κόσμο αφορά την ε, ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, επικεντρώνεται όμως αποκλειστικά και μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτι που δεν ισχύει για το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020. Θα διοργανώσουμε ένα εργαστήριο, ένα workshop, μια, ένα σεμινάριο για το θέμα αυτό και ίσως θέλουμε και ένα ειδικό σεμινάριο για τις επιδόσεις του ΣΥΠ και την διεθνοποίηση του κόσμου και το θέμα του διοικητικού άχθους. Δεν θα ήθελα τώρα να μακρηγορήσω. Θα ευχαριστήσω τους ομιλητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα σχόλιά τους και σας διαβεβαιώ ότι κατά τη γνώμη μου θα διαμορφώσουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα για να συμπληρώσουμε τις ε, υπάρχουσες δυνατότητες και προσπάθειές μας. Κύριε Λάγκεν, δεν ξεκινούμε εκ του μηδενός. Δίκιο έχετε ότι θέλουμε να έχουμε καλύτερες ε, επιδόσεις και πολύ περισσότερες προσπάθειες. Από τον κύριο Μπάγκεμαν, από τη θητεία του κύριου Μπάγκεμαν, πολλά έχουν γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2008 είχαμε το Small Business Act και το 2011 είχαμε την αναθεώρηση του Small Business Act. Είχαμε το έρασμος για τους νεαρούς επιχειρηματίες. Είχαμε τις ε, οικογενειακές επιχειρήσεις, την απλούστευση της χρημα τους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς, την διεθνοποίηση. Έχουμε πολύ περισσότερες ε, προσπάθειες που έχουν γίνει από την εποχή του κ. Μπάγκεμαν. Αν δεν πίστευα σε όλες αυτές τις πρόοδους και στις ε, προσπάθειες, δεν θα ήμουν στη θέση που είμαι. Σας ευχαριστώ πολύ και να πω ότι η πρόεδρος θεώρησε ότι είμαι ο πρεσβύτερος, ο, ο ε, ίσως ε, δεν ξέρω λόγω ηλικίας, αλλά εν περιπτώσει ο κύριος Λάγκεν έχει το λόγο. Μία ερώτηση έχω να κάνω προς τον κύριο Γενικό Διευθυντή. Το ερώτημα που έθεσαν πολλοί σε ό,τι αφορά τη διάκριση μεταξύ των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε δηλαδή αν θα ελεγχθούν επιτέλους οι ορισμοί. Ναι, απάντηση. Νομίζω ότι σας απάντησα ότι θα γίνει μία μελέτη για τους ορισμούς, αλλά για να είμαστε σαφείς, ε, να είμαι σαφείς, κύριε Λάγκε, δεν θέλω να ξοδέψω χρόνια να συζητάω ορισμούς και στο μεταξύ να μην κάνουμε τίποτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλή και οι ορισμοί, αλλά ακόμα καλύτερα το να δράσουμε. Και όπως σωστά τονίστηκε, υπάρχει μια αίσθηση κατεπήγοντος. Ξέρω ότι όλοι, σε όλους αρέσουν οι ορισμοί. Και το να συμφωνήσουν 27 χώρες και όλοι οι βουλευτές επί ενός ορισμού δεν πρόκειται να επιτευχθεί γρήγορα. Και στο μεταξύ τι θα κάνουμε με τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Κούκοβιτς ότι υπάρχει μια αίσθηση κατεπήγοντος. Θα γίνει η μελέτη, θα γίνει η συζήτηση για τους ορισμούς, αλλά δεν πρόκειται στο μεταξύ να αναστείλουμε την πρόοδο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι να συμφωνήσουμε για τον ορισμό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. 11 Απριλίου το εργαστήριο για τα χρηματοπιστωτικά ε, μέσα και στις 25 για το σεμινάριο για την συμφωνή, ε, συμμετοχή του προγράμματος SIP. Θα συζητηθούν θέματα ευελιξίας. και ανοίγματο των ε, προγραμμάτων, γιατί ξέρω ότι πολλοί απορρίπτονται σε τελική ανάλυση και περνάμε τώρα στο πέντο σημείο της ημερίας, της διάταξης ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα και εμπορικές πρακτικές. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον συνάδελφο Ρούμπιχ που είναι εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα αυτό εντάσσεται και στην, στην ίδια προβληματική. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για τις διεθνείς ε, προδιαγραφές και προϋποθέσεις ε, και πώς μπορούν να βελτιωθούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ και πολύ, εδώ πολλά χρόνια στον ΠΟΑ γίνονται παρόμοιες συζητήσεις και μιλάμε καταρχάς για τις εμπορικές διευκολύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως θα πρέπει το θέμα αυτό να το επεξεργαστούμε ξεχωριστά για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και να ζητήσουμε στην Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Χρειαζόμαστε και μητρό στον ΠΟ για όλους, όλους τους δομευτικούς όρους εισαγωγής και εξαγωγής, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε το μίσο που επικρατεί μεγάλη διαφθορά, να διαπιστώσουν τι είναι πραγματικά δεσμευτικό σε ό,τι αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να οριστούν, ε, να υπάρξει διαφάνεια. Ο δεύτερος τομέας είναι ε, τα χρηματοοικονομικά, όπως και στο πρόγραμμα COSME. Χρειάζονται πόροι για τις εγγυήσεις, χρειάζονται ήπια δάνεια, χρειάζεται ένα σενάριο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μας, γιατί φυσικά εδώ ε, μιλάμε σε μεγάλο ποσοστό για κεφάλαιο κινδύνου και η συγχρηματοδότηση αυτού του κεφαλαίου αποτελεί μια πραγματική πρόκληση. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία. Το τρίτο θέμα είναι η υπεραιτέρω κατάρτιση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό κλάδο ασφαλώς, ε, κυρίως δεν έχουμε αρκετούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, αλλά και αρχές ε, και υπηρεσίες ε, παροχής συμβουλών σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτή τη διαφύγη των εγκεφάλων, σε αυτό το brain drain που επικρατεί. Και θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί φυσικά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ πολιτισμών και ανάλογα να ε, οδηγήσει σε καλές επαφές. Τέταρτον, το πρόγραμμα Εράσμου για Νεαρούς Επιχειρηματίες θα πρέπει να διευρυνθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το Εράσμου Μούντου, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα στο οποίο οι νέοι επιχειρηματίες θα κάνουν ανταλλαγές και εντός της Ευρώπης αλλά και με άλλες υπήρους και έτσι θα λάβουν κινήτρα για να επισκεφθούν ενδεχομένως προμηθευτές, πελάτες. Αυτό νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει και τον σκοπό Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη καινούργια ε, υπηρεσία εξωτερική δράσης. Ε, κατά πέμπτον, σε ό,τι αφορά την τεχνική αρρωγή, σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία. Αυτό αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κλάστερ καταρχά και δίκτυα όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να αναλύσουμε τι γίνεται και σε άλλες επίρους. Να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Να αναπτύξουμε benchmarks και ένα scoreboard ενδεχομένως για να αποφασίσουμε τελικά ποιο είναι το καλύτερο πρόγραμμα για την Ευρώπη. Να κοιτάξουμε τι γίνεται στις περιφέρειες στα κρατημέλη, στις πόλεις. Θα μπορούσαν να υπάρχουν, για παράδειγμα, συνεργασίες μεταξύ πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο και να υποστηριχθούν για τη δημιουργία επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων. Θα μπορούσε να υπάρξει περιφερειακή δικτύωση και των περιφερειών. Πολλέ δραστηριότητε μπορούμε να φανταστούμε και νομίζω ότι δικό μα καθήκον είναι να θέσουμε τα νέα σημεία προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ρούμπιχ. Και τώρα θα περάσουμε στους σκιώδεις εισηγητές. Θα πω τα ονόματά τους και όποιος είναι από. Αν θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος ε, συνάδελφος, η κυρία Τόγια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Θα το αναλάβετε εσείς. Έχετε το λόγο. Αν θέλετε να μιλήσετε για την κυρία Τόγια εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών, παρακαλώ πάρτε το λόγο. Κυρία Χέρτσοκ, όχι. Πριν από λίγο είχα μιλήσει εκ μέρους και όδους Όταν έλαβα προηγουμένως το λόγο, εξέφρασα την σκέψη και της τη ηγετριάς μας. Ο κύριος Γιώχανσον απουσιάζει. Ο κύριος Μπιουτικόφερ επίσης απουσιάζει. Η κυρία Φόρτ από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Και μετά θα δούμε ποιοι εκπρόσωποι των άλλων ομάδων θέλουν το λόγο. Κυρία Φόρτ, δικαιώστε το λόγο θέλετε. Αργότερα θα προτιμούσα κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Ωραία, τότε ποιος θέλει το λόγο για την έκθεση του κυρίου Ρούμπιχ. Yeah, you have the floor. Yes? Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν συνεννοηθήκαμε. Ε, δεν θα ήθελα να εκπροσωπήσω εδώ κάποιον άλλον ή κάποιο και οδησηγητή, απλώς ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη. Πειράζει? Τι γίνεται καταρχήν με το μέγεθος των επιχειρήσεων έχουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις μικρές και τις μεσαίες. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες, οι τύποι των υπηρεσιών που έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερων εξαγωγών και τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν σε τεχνολογικές πλατφόρμες και σε διάφορα δίκτυα γιατί τα δίκτυα και οι πλατφόρμες είναι μια καλή ευκαιρία για την ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία, ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. vielen Dank. Äh, Mr. you have the floor. Καλώς. Κύριε Πυρίγιο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πυρίλο, μάλλον. Και μετά, κύριε Φόρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ρωτήσατε για τη γνώμη της κυρία Στόγια που είναι η σκιώδη συγκήτριά μας, αλλά στην προηγούμενη συζήτηση έλαβε το λόγο και μας μετέφερε την γνώμη της κυρία Στόγια η κυρία Χέρτσοκ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την έκθεση του κυρίου Ρούμπικ. Θα ήθελα να το συγχαρώ για την έκθεση του και για τα σχόλιά του. Και πάνω απ' όλα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις προάλλες στην Ολομέλεια είχαμε μια ψηφοφορία για την ε, ταχύτερη ε, ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Αλληλευτικού Ταμείου. Και αυξήσαμε την ε, κοινωτική χρηματοδότηση από το 10% ακριβώ επειδή έχουμε πολλέ μικρέ και μικρομεσαίε επιχειρήσει που δεν είναι σήμερα σε θέση να απορροφήσουν τα κονδύλια που δικαιούνται γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη δική τους χρηματοδότηση για να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες. Διανύουμε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι πραγματικά ο νοτιός μυαλός, ο σκελετός του ε, οικονομικού και του βιομηχανικού ιστού και του έθνους. Αν θέλουμε να αναπτυχθεί και να διαβριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει το know-how, η τεχνογνωσία που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια χώρα να μπορεί να ε, μεταλαπαθευτεί και σε άλλη χώρα. Γιατί υπάρχουν χώρε στις οποίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι πιο προηγμένε, ενώ σε άλλε έχουν μείνει πιο πίσω. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε τη μεταβίβαση τεχνογνωσία από τη μια χώρα στην άλλη, από τι επιχειρήσει μικρομεσαίες μια χώρα προ τι μικρομεσαίες επιχειρήσει μια άλλη. Τώρα, υπάρχει πρόβλημα με... Υπάρχει πρόβλημα του σπόρου. Δυστυχώ υπάρχει μια μεγάλη σπάνη σπόρων, αν και σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν περισσότερο από ποτέ να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Και το θέμα της κατάρτισης, ε, μας είπε προηγουμένως ε, ε, πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα ο Γενικός Διευθυντής. Μίλησε για συγχρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων και από άλλα ταμεία, όπως είναι το Κοινωνικό Ταμείο, το Περιφερειακό Ταμείο. Η έκθεση πάντως που πρόκειται να ψηφίσουμε θα πρέπει να λάβει υπόψη και τον ορίζοντα 2020 και να, το, να συνδυάσουμε αυτά τα κονδύλια με τις πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που επαναλαμβάνω σήμερα δεν είναι σε θέση περισσότερες να συνεχίσουν την επιβίωσή τους στην αγορά εξαιτία αυτού του κατακαιρματισμού τη ενιαία αγορά, που πραγματικά δεν είναι ενιαία, αλλά είναι κατακαιρματισμένη. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιόρτ. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κανένα δύο σχόλια κύριε Πρόεδρε σε αυτά που αναφέρθηκαν από τις διανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ένα αφορά την ενημέρωση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι δύσκολο και ακούω συχνά παράπονα ότι είναι τόσο πολλά τα γραφεία ενημέρωσης, είναι τόσο τόση μεγάλη πληθώρα των πληροφοριών που στο τέλο ε, πελαγώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που πραγματικά χρειάζονται. Καταλαβαίνω λοιπόν την επιθυμία τη ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλούστευση. Καλό θα ήταν να απλουστευτεί βέβαια και η κυβερνητική δομή για να αποφευθούν οι επικαλύψει θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ήδη υπάρχ, τα ήδη υπάρχοντα γραφεία και τα helpdesk λειτουργούν, ώστε να μην προσθέτουμε σε αυτή τη σωρία των πληροφοριών. Το θέμα είναι να είναι οι αποτελεσματικέ πληροφορίε που υπάρχουν και όχι να υπάρχουν άπειρε πληροφορίε αναποτελεσματικέ. Και το θέμα της ε, συνδρομής, της εμπορικής συνδρομής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόσβαση στις χώρες BRICS ήταν πολύ σημαντικό. Να διδαχθούμε από τις χώρες που έχουν καλύτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τους όλες. Έτσι ε, θα έχουμε και παροχή πιο ακριβών και σωστών πληροφοριών. Το θέμα των υπερημεριών ε, πληρωμών. Είχαμε την οδηγία για τις υπερήμερες πληρωμές από πολλέ απόψει είναι θετική αυτή η οδηγία, αλλά είναι επίση ε, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα οδηγία που είναι στα χαρτιά καταπληκτική, αλλά τα αποτελέσματά της δεν είναι ομοιόμορφα. Άκουσα από μια μεγάλη ε, επιχείρηση που σταμάτησε να χρησιμοποιεί ως προμηθευτέ μικρομεσαίες επιχειρήσει εξαιτία οδηγία για τις υπερήμερες ε, πληρωμές. και επίσης επιχειρήσεις αφήνουν τα προϊόντα στις, στα ράφια τους πολύ πολλά χρόνια και έχουν προβλήματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη ροή των μετρητών. Δυστυχώς ήταν ε, στα χαρτιά καλή η οδηγία για τις υπερήμενε ε, πληρωμές, αλλά στην πράξη ε, επιδίνωσε την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντί να τις βοηθήσει όπως ήταν αρχικά ο στόχος της. Θα πρέπει λοιπόν όταν ανακύπτουν προβλήματα με τις οδηγίες να τα εξετάζουμε. Τι μιλάτε για την με ενσωμάτωση τη οδηγία των υπερήμερων πληρωμών στην εθνική νομοθεσία. Γιατί νομίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία ήδη την έχει ε, ενσωματώσει. Πού υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω ότι η Γαλλία ε, υιοθέτησε ακόμη βραχύτερε προθεσμίε από ό,τι οδηγεί και εκεί δημιουργήθηκαν προβλήματα με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Καλώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει κάποιε απαντήσει, αν το επιθυμεί, και ε, στη συνέχεια για να ανακεφαλαιώσει στον εισηγητή μα τον κύριο Ρούμπιχ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ λακωνικό, γιατί νομίζω ότι καλύψαμε στην προηγούμενη συζήτηση τα περισσότερα από τα θέματα αυτά. Θα ήθελα απλώ να πω ότι χαίρομαι για την έκθεση του κυρίου Ρούμπιχ. Πιστεύω ότι θα παρουσιάσει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κέρια ζητήματα που ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως είναι διεθνοποίηση, βιομηχανική πολιτική, ε, ρύθμιση αγοράς. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρουμπιχ που είναι πολύ σημαντικό σύμμαχός μας στον αγώνα που θέλουμε να δώσουμε υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε απογραφή των ε, διατάξεων του ΠΟΕ, soft law, προσόντα, έρασμος για τις νέες επιχειρήσεις, προδιαγραφές, ε, θύλακες αριστείας, ε, δίκτυα. Όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να καλυφθούν και από το κόσμο και από το ΣΥΠ. Και σας ευχαριστώ γιατί είναι πραγματικά σημαντικές προτεραιότητες. Ε, σε ό,τι αφορά κάποια ζητήματα που θίξατε, θα ήθελα να πω ότι αντιλαμβανόμαστε τα, τα προβλήματα ενημέρωση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που έθιξε η κυρία Φόρτ. Και θα πρέπει να αποφύγουμε να κατακλείζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πληθώρα πληροφοριών που σε τελική ανάλυση δεν τους ε, βοηθούν. Γιατί μπορούμε να πνίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμη και με αυτόν τον καταιγισμό από πληροφορίες που τελικά δεν μπορούν να αξιοποιήσουν. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας ε, των χωρών μέλων, ήδη προσπαθούμε να κάνουμε έναν απολογισμό των διαφόρων επιδόσεων για να εκμεταλλευτούμε τις καλύτερες. Ο Αντιπρόεδρος Σταγιάννη έχει στείλει επιστολή σε όλες τις χώρες και η οδηγία αυτή θα πρέπει να τεθεί ε, σε ισχύ μέχρι τις 15 Μαρτίου του 2013. Οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να καταβάλουν τα χρέη τους μέσα σε 30 μέρες. Ο κύριος Σταγιάννη έστειλε επιστολή σε όλες τις χώρες και είπε μην περιμένετε το Μάρτιο του 2013. Σπεύστε, γιατί το πρόβλημα που έχουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ότι δεν έχουν ε, προ... δεν είναι ότι έχουν πρόβλημα πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είναι ότι γίνονται οι τραπεζίτες των τοπικών, ε, της τοπικής αυτοδίκης που δεν πληρώνει τα χρέη της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε μόνο να εξασφαλίσουμε πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο δανεισμό, αλλά και εμπρόθεσμη αποπληρωμή των χρεών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μην αναγκάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνονται τραπεζίτες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μερικές χώρες όπως η Ολλανδία ήδη ενημέρωσαν ότι θα εφαρμόσουν την οδηγία πολύ πιο σύντομα από την ε, πρόβλεψή της για τη θέση ισχύ, την καταληκτική της προθεσμίας. Ό,τι αφορά τον κύριο Πυρίλο, συμφωνώ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο σκελετός, ο μυελός της οικονομίας και θα πρέπει ε, να φροντίσουμε όλοι οι μηχανισμοί να ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση και σα διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει τις προτάσεις και τις τάσει. Θέλουμε οι μηχανισμοί και τα εργαλεία μας ε, να στηρίζουν την πολιτική μας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι προτάσει για τα προσόντα, του πόλου αριστείας, ε, τη πρόσβαση ε, στο δανεισμό και στο κεφάλαιο, η αξιοποίηση και η ανταλλαγή των εμπειριών. Όλε αυτέ οι προτάσει είναι χρήσιμε και θα τι λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ κύριε Σουρεμπίχη. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γενικό Διευθυντή γιατί θεωρώ ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα του Επιτρόπου Τατζάνη, θέτει τις γενικές ε, συνθήκες και όρους πλαίσιο και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για το πώς θα καταφέρουμε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας ε, που είναι διεθνείς προκειμένου μέσω του διαδικτύου μέσω της ε, παγκόσμιας επιμελητίας που έχει προκύψει. Πώς θα καταφέρουμε λοιπόν να τις τοποθετήσουμε με σωστό τρόπο στο διεθνή ανταγωνισμό. προκειμένου να δραστηριοποιηθούν, για παράδειγμα, σε μια νέα ήπειρο. Και γι' αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι το πρόγραμμα Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες ε, αποτελεί μια πολύ καλή προσέγγιση. Θα πρέπει να θέσουμε ένα στόχο και θα μπορούσαμε να μάθουμε και να ενταχθούμε και από τους Κινέζους, βλέποντας πόσους νέους στέλνουν στο εξωτερικό. Στη Σαουδική Αραβία, 8 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά και να ενταχθούμε πολλά από άλλες χώρες του κόσμου. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να τονωθεί ιδιαίτερα και νομίζω ότι πρόκειται για έναν τομέα όπου μπορούμε να απευθυνθούμε στους νέους και μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όταν μιλάμε για 23 εκατομμύρια ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη, μα κάθε επιχείρηση έναν εργαζόμενο παραπάνω να έπαιρνε, δεν θα υπήρχε ενεργεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά πολύ καινούργιο το δυναμικό αυτό που έχουν να προσφέρουν ιδιαίτερα οι νεαροί επιχειρηματίε. Να ευχαριστήσω και του συναδέλφου, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε να σκεφτούμε. Γιατί μπορούμε να έχουμε επιτυχία μόνο αν προσφέρουμε υπηρεσίε και προϊόντα τα οποία θα αγοράζονται τελικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί το στόχο μα, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε και την κρίση του χρέου των ευρωπαϊκών κρατών. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, στο 6, ανάπτυξη τη συνεργασία με του πέραν των συνόρων μία μας εταιρούς στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, στρατηγική προσέγγιση ενός ασφαλούς, βιώσιμου και ανταγωνιστικού ενεργειακού εφοδιασμού. Να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Χέρτσογκ. Έχετε το λόγο, κυρία Χέρτσογκ. She's phoning. Α, παίρνει τηλέφωνο. Μιλάει στο τηλέφωνο. Frau Kollegin Herzog, Miss Herzog. Κυρία Χέρτσοκ, λέει ο πρόεδρο. Έχετε το λόγο για το επόμενο θέμα μα. Είστε η συγγήτρια για το 6. Για το 6. Έχετε το λόγο. Μπορείτε να μα μιλήσετε. Κύριε Κρότσμαν, συμπαθάτε με. με πήρε συνεργάτη εδώ για κάτι πάρα πολύ επίγον. Κύριε συνάδελφοι, πάντως, ε, όσον αφορά τις τροπολογίες για την έκθεση που αφορά την εξωτερική πολιτική ενεργείας, σας ενημερώνω ότι δυστυχώς ή δυστυχώς η ΑΦΕΤ ακόμα δεν έχει τελειώσει το δικό της κείμενο. Επομένως, η δική μας 7 ή 8 Μαΐου θα ψηφιστεί. Με τη μέρα της Ευρώπης και επομένως έχουμε το χρόνο για σας επίσης. Σας ευχαριστώ όσον αφορά όλες αυτές τις τροπολογίες. 182 μου έχετε υποβάλει. Οπότε θα προσπαθήσω να φτιάξουμε όσο γίνεται περισσότερες συμβαστικές. Συνάδελφοι, οι περισσότεροι κατατείνονται στην ίδια κατεύθυνση. Προς εκείνη στην οποία κινούμε και εγώ. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για τους χιώδεις ηγετές. Ευχαριστώ. Καρβάλιο, Τούρμες και τους άλλους, Βάλεν και λοιπά. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη φάση δεν χρειάζονται περισσότερα, διότι δεν έχουμε θέματα ιδιαίτερα. Άρα να ψάξουμε μέσω συμβαστικής να βρούμε το καλύτερο κείμενο. θέλουμε να βρούμε μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά. Να έχουμε καλύτερο συντονισμό και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα έχει ενιαία φωνή πάνω στο θέμα. Πάντως νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πιο ενδιαφέρον έχει η γνώμη των συναδέλφων για τα καθεσία μου παρά η δική μου άποψη. Ευχαριστώ να παρακαλέσω τους όντες εισηγητές να ε, μας παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε τρία μόνο λεπτά γιατί στις ε, πέντε θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Από το ΕΛΚ, η κυρία Καρβάλιο. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Χέρτσοκ. Επιτέλεσε έργο αξιόλογο. Συγενικές συμφωνώ με τα όσα μας ανέπτυξε. Επίσης, Νομίζω ότι με αυτή την έκθεση υποστηρίζουμε το νομοθετικό έργο ε, και το έδαφος το οποίο προλύωνε κύριε Κάνης. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει με τις τροπολογίες να βελτιώσουμε διάφορα σημεία όπω ε, όπως ας πούμε την ε, ισορροπία μεταξύ καταναλωτών παραγωγών, ζήτησης προσφοράς μεταξύ αναδυόμενων χωρών, βιομηχανικά προηγμένων, να συγκεράσουμε τις επιθυμίες, τις ανάγκες Βορρά, Νότου, Ανατολής, Δύσης, Ατλαντικού, Μεσογείου και έτσι να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Δηλαδή να έχουμε ποικιλία για τις χώρες διέλευσης και τις χώρες προέλευσης. Να δούμε τι θα γίνει με την ε, συνεργασία, την τεχνολογική έμφαση όσον αφορά τα πρότυπα, την ανάπτυξη νέων προτύπων και στάνταρ, όπως λέμε. Επίσης, δεν διαπιστώνω να υπάρχει κανένα πρόβλημα, να υπάρχει κανός είδους διαφωνία σε σχέση με τις υποβληθήσεις τροπολογίες. Οπότε, Νομίζω στην επόμενη φάση θα έχουμε αρμονική συνεργασία και με ομαλό τρόπο να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές. Και σας ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ και τώρα για την εβδομάδα του Άλντε, κύριος δεν είναι εδώ κανείς, αλλά ο κύριος Τούρμες για τους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Μάλλον έτσι είναι ευκολότερο να με καταλάβει και η Edith. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κείμενό σου. Το ε, βασικό θέμα είναι αυτό το οποίο τόνισε και εσύ. Να υπάρχει περισσότερο κρατών μελών και να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη ενημέρωση, πληροφόρηση για τις πολιτικές αυτές με την Ινδία, με την Κίνα, τι γίνεται με τις διεθνείς φορείς όπως ε, τη Διεθνή Υπηρεσία Ενεργείας γιατί έχουμε εκεί πολυφωνία όσον αφορά την εκπροσώπηση τη Ένωση από διάφορα Χρειάζεται περισσότερο συντονισμό. Τώρα, όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία για τεχνολογία και τι θα γίνει με του εταίρου μα, θα πρέπει καλύτερα να εξετάσουμε το τι ισχύει όσον αφορά τις επόμενες δύο δεκαετίες τις αγορές, τον όγκο των εμπορικών ροών και έτσι να κάτσουμε και να κάνουμε μια εκτίμηση καλύτερη. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω πάντως η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, οι νόσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, η διαβίβαση, η μεταφορά, τα μικροδίκτυα. Μιλάμε για 75-80% αν όχι περισσότερο από τον όγκο της ενέργειας που τίθεται σε εμπορία. και όλα αυτά τα δις που έχουμε δεσμεύσει μέσω του προπολογισμού δεν έχουν βοηθήσει πολύ. Άρα να λάβουμε υπόψη τι θέλει η αγορά, πώς θα πάει η αγορά για τα δίκτυα και για τις μας. Τώρα, τα θέματα ανάπτυξης, να προσέξουμε περισσότερο το ότι φέτος Ο ΕΕ είπε ότι είναι η χρονιά τη καλύτερη πρόσβαση στην ενέργεια. Έχουμε την εκδήλωση που οργάνωσε για τον Απρίλιο ο Μπανκιμών. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί η διαδικασία του Ρίο, η διαδικασία δική μας, αν θα συγχωνευτούν, τι θα ισχύσει. Όμως μας δίνεται μοναδική ευκαιρία φέτος για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θέλουν με εθνικά προγράμματα να προχωρήσουν για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας και εμείς αντίστοιχα να έχουμε προβλέψει τον προπολογισμό, τεχνική αρρωγή, ελάχιστα πρότυπα, ετικετοποίηση, ετικετοθεσία. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας όπου μπορούμε να συνεργαστούμε να ενώσουμε τις προσπαθειές μας τώρα σαν φορά τα βιοκαύσιμα. Κατά πάσα πιθανότητα σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει κάποιες προτάσεις για τη χρήση της γης, πώς όλα αυτά θα γίνουν λειτουργικά μέσω του κοινοτικού δικαίου γιατί αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τις εξαγωγικές αγορές και να βοηθήσουμε την εξαγωγή από τι αντισώμενε χώρε προς εμάς, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα βιοκαύσιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τι θα κάνουμε με αυτό. Τι είναι με τις περιφερειακές αγορές. Οι παλέτες, λέει ο μιλητής, προέρχονται από την Ευρώπη, ό,τι έχουμε σήμερα. Όμως, πάρα πολύ. Σφαιρίδια, σφαιρίδια εννοεί. Ρωσία, Γκάνα, προέρχονται από, από παντού. Αφρικανικές χώρες, άλλε πέραν τη Γκάνας. Άρα υπάρχει μια παγκόσμια αγορά για την βιομάζα. Όμως, εάν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε αγορές και να μην είναι πάνω κάτω η κατάσταση, on-off, θα πρέπει να έχουμε κάποια κριτήρια βιώσιμα ή κριτήρια βιωσιμότητας και να βοηθήσουμε τι ανθρώπινε χώρες να αναπτύξουν, να εκμεταλλευτούν τι δυνατότητέ του και όχι μόνο να θεσπίζουν νομοθεσία αλλά και την εφαρμόζουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Edit. Ήταν μια εξαιρετική πράγματι ε, αναφορά κυρία Χέρτζοκ πολύ καλογραμμένη και πολύ λίγα είναι αυτά τα οποία θα μπορούμε να προσθέσουμε. Ε, στην αναφορά είναι δύο-τρία σημεία που θα ήθελα να αναδείξω. Στην αναφορά σας φαίνεται η τεχνογνωσία σας για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα δύναμο κομμάτι που αφορά την, νότιο, την νότια και ανατολική Ευρώπη, νότια-ανατολική Ευρώπη, όπου εκεί έχουμε αρκετές εξελίξεις στην ενέργεια. Γι' αυτό έχω κάνει α, κάποιες ε, προτάσεις, προσθήκες που να αναδείξουν ε, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά, στο Νότο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ε, μία άλλη, ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι εμφανές στην ε, αναφορά της κυρίας Χέρτζοκ ότι έχει κατά νου πάντα το θέμα του μονοπωλίου ή της μονοπωλιακής ε, συνεργασίας της Ευρώπης με τη Ρωσία. Η πρότασή μου είναι ότι με τη Ρωσία θα πρέπει να μπούμε σε ένα διάλογο που να προσδιορίζει δημιουργικά και αμοιβαία αποδεκτά μέτρα τα οποία θα αποσκοπούν στη μείωση των διαφορών των αποκλήσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο αγορών ενέργειας της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη ρωσική αγορά. Οπότε έχω κάνει ένα amendment και από αυτού του θέματος. Επίσης αναφέρομαι στο shale gas γιατί υπάρχει μια προσπάθεια του Κλοντ να μην αναφέρεται μέσα. Είδα ότι ζητάει ο Κλοντ ε, ε, να κάνουμε delete το θέμα του shale Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ένα καινούριο προϊόν το οποίο βγαίνει στην παγκόσμια αγορά, υπάρχει σε τρίτες χώρες, έχει αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της Αμερικής και έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων στον πλανήτη οπότε μία αναφορά στο shale gas κακό δεν κάνει. Δεν αναφερόμαστε περιβαλλοντικά ή οτιδήποτε αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτό το οποίο αναφέρεται ως προϊόν που συνεργαζόμαστε με τις τρίτες χώρες. Κλείνοντας επισημένο, οι σχέσεις στον τομέα της ενέργειας απαιτούν προβλεψιμότητα, σταθερότητα και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Γι' αυτό πρέπει πάντα να προσέχουμε να μην αναμειγνύουμε εξωτερικές σχέσεις με την ενεργειακή επάρκεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Τρικαστήγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις τροπολογίες μου, γιατί στις 5 κανονικά πρέπει να είχαν αρχίσει οι συντονιστές στη συνεδριασή τους, ήδη είναι 5 και 5, γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο. Κύριος Βινταλ Κουάδρας. Ευχαριστώ. Η έκθεση της κυρίας Χέρτσοκ είναι συμπληρωματική της έκθεσης Κάρνς για τους μηχανισμούς ανταλλαγής ε, πληροφοριών σε ό,τι αφορά διακυβερνητικέ συμφωνίε με τρίτε χώρε για ενεργειακά ζητήματα. Θεωρώ ότι αυτέ οι δύο εκθέσει αποτελούν ε, τις... δημιουργούν ένα σύνολο που μας επιτρέπει να δώσουμε μια όθηση για την ανάπτυξη μιας γνήσιας εξωτερικής ευρωπαϊκής πολιτικής για ενεργειακά θέματα. Μια τέτοια εξωτερική ενεργειακή πολιτική θα πρέπει αναφυσβήτητα να αποτελέσει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επισημαίνει άλλωστε και η εισηγήτρια με πολύ εύστοχο τρόπο. Μας λέει σε κάποιο σημείο ότι η τεράστια μας εξάρτηση σε ό,τι αφορά την προμήθεια ενέργειας ε, δημιουργεί ε, μια δυναμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την δυναμία μας θα πρέπει να τη μετατρέψουμε σε ισχύ, γιατί χάρη σε αυτή την εξάρτηση είμαστε ο μεγαλύτερος αγωγές ενέργειας. Και αν μιλούμε με ενιαία φωνή, αυτή την, το τρωτό μας σημείο, αυτή την αδυναμία μας θα τη μετατρέψουμε σε ισχύ, σε δύναμη. Και αυτό θα πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε, συνενώνοντας τις φωνές μας και με συσπήρωση. Αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Το σχέδιο έκθεση κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ισορροπημένο και πολύ εύστοχο. Έχει κάποια σημεία που με βρίσκουν πλήρως σύμφωνο. Για παράδειγμα, η μνήα της ε, σημασίας που έχει μια πλήρως ολοκληρωμένη ενεργειακή εσωτερική αγορά, που είναι πολύ σημαντικό σημείο για να έχουμε μια πραγματική ενεργειακή διπλωματία επιτυχημένη, ή το σημείο που λέει ότι μόνο η διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση η και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μπορούν να αντισταθμίσουν την αυξανόμενη εξάρτησή μας από τρίτες χώρες. Μία τόσο καλή έκθεση <laughs> είναι δύσκολο να τροποποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, με, με ε, πολύ μετριοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη προσπάθησα να συμβάλλω στη βελτίωση έκθεση μετροπολογία, για παράδειγμα για τη βελτίωση της, του εσωτερικού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου ε, στις, στα διεθνή φόρα και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις να υιοθετείται κοινή θέση των κρατών μελών για ενεργειακά θέματα. Επιμένω στην ανάγκη εκπόνησης μιας στρατηγικής απέναντι σε χώρες που αυξάνεται ε, με ταχύτητα ρυθμούς η ενεργειακή του κατανάλωση γιατί πρόκειται για αναδυόμενες οικονομίες με πολύ σημαντικούς ε, ρυθμούς ανάπτυξης ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες αυτές λοιπόν Επίσης, ε, πιστεύω ότι η ενέργεια θα πρέπει να αποτελέσει κέριο σημείο και των αναπτυξιακών μα πολιτικών. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα τα συμπεριλάβω σε τροπολογίες που ελπίζω ότι θα γίνουν δεκτές από την εισηγήτρια ως θετικές ε, πινελιές στην έκθεσή της. Ευχαριστώ πάντως την εισηγήτρια και τη συγχαίρω για την καταπληκτική της έκθεση. Ο κύριος Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, να είστε σύντομο, κύριε Οντή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα μικρό πρόβλημα μετάφραση. Στην παράγραφο 20, εκεί που αναφέρονται τα πυρηνικά θέματα, η ασφάλεια, το σιωχτέ, το safety στα αγγλικά έχει μεταφραστεί στο security, ασφάλεια. Η προστασία στα αγγλικά έχει μεταφραστεί σε ασφάλεια. Γιατί η η ασφάλεια είναι θέμα κοινοτικό, η προστασία είναι θέμα εθνικό. Σε ό,τι αφορά μια πολύ παλιά ιδέα του Ζακ τελόρ και που ακούγεται όλο και πιο συχνά το τελευταίο χρόνο για την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας. Είναι καλή αυτή η ιδέα τελικά ή όχι. Θα ήθελα επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μία σύγκριση παγκόσμια. Να δούμε οι άλλοι πυροί με τις οποίες έχουμε ανταγωνισμό, πώς διαχειρίζονται τα προβλήματα ε, ενεργειακής ε, ε, εξασφάλισης του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Γιατί όλες οι πυροί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση για να δούμε αν πραγματικά έχει νόημα μία ευρωπαϊκή κοινότητα ενέργειας. Παρακαλώ, ακούσατε κυρία Μάρκες τις ερωτήσεις του κυρίου Οντή. Μπορεί να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, και ευχαριστούμε και για τις τροπολογίες που υποβάλλατε. Με αυτές αναγνωρίζετε το πόσο σημαντική είναι η εξωτερική ενεργειακή πολιτική για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της Ένωσης. Επίσης, έτσι καταδεικνύεται ότι χρειάζεται να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τις επαφές μας με τους διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ισορροπία, κάτι το οποίο το πετυχαίνουν οι τροπολογίες και με εταίρους και με ανταγωνιστές, να δούμε τι θα κάνουν. Οπότε, αν μου επιτρέπετε θέλω να σας αναφέρω άλλα δύο σημεία. Για την ενεργειακή κοινότητα. Να διευκρινίσουμε ότι όσον αφορά τη σχετική πρόταση για το νομοθέτημα για κάποιο είδους παρατηρητήριο, όπως γνωρίζετε, ήδη έχουμε ένα σύστημα παρατήρησης αγοράς. Από το 2008 λειτουργεί. Υπάρχει σχετική αποστολή. Μαζεύουμε πληροφορίες, αναλύουμε τις αγορές, και έτσι βοηθούνται αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Δημοσιεύσεις σε τακτά διαστήματα μελέτες έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ένα άλλο είναι το ότι στην ε, ανακοίνωσή μας είπαμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε ένα νέο ρόλο όσον αφορά τις ε, συνθήκες με τις ε, άλλες χώρες. Ο σκοπός είναι να διευκολύνονται οι υποδομές μεγάλης κλίμακας, ρυθμιστικά θέματα και άλλα. Όχι, όχι, δεν ασχολούμαστε με τον όγκο των ροών, ούτε την τιμολογιακή πολιτική. Αυτό αλλού ρυθμίζεται, στους εμπορικούς χώρους, εμπορικά κέντρα. Όσον αφορά την ε, ενεργειακή κοινότητα, η ανάπτυξη μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής είναι μια διαδικασία που προχωράει βαθμία. Σε αυτή τη φάση δεν απαιτούνται νέες θεσμικές ρυθμίσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πολλά για να εξευρωπαϊστεί η δική μας πολιτική. Και υπάρχει μια νέα έκθεση όσον αφορά την περαιτέρω δράση σχετικά με αυτό και αυτό περιλαμβάνει και την εξωτερική πτυχή. Επίσης, πάρα πολλές επιστροπολογίες θίγουν ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά με εξωτερική πολιτική ενέργεια πολιτική υποδομής, Αυτά θίγονται σε ειδικέ εκθέσεις, χωρίς να προδικάζουμε το ότι εσεί θα κρίνετε σχετικά. Και σας ευχαριστώ. For the, for summary. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Χέρτσοκ, θέλετε να δευτερολογήσετε, να συνοψίσετε. Ναι, ναι, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να σας πω με λίγα λόγια ότι... Όντω. στο ίδιο μήκο κύματος κινούμεθα, εγώ και οι τροπολογίε. δεν εκπροσωπεί μόνο την πλευρά της ζήτησης, αλλά και της προσφοράς. Ιδίως για τις νέες τεχνολογίες και τη μεταφορά γνώσης και Επίσης έχουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία, άρα και αυτό πρέπει να το δούμε. Στους επόμενους μήνες θα βελτιώσουμε το κείμενο με τροπολογίε. Να κάτσουμε να δούμε τι βέβαια θα πει, γιατί τους περιμένουμε σε σχέση με όλα τα θέματα τα σχετικά με τους διεθνείς συνομιλητέ μας. Και άλλες αρμόδιες επιτροπέ όπως η ΝΤΕΒΕ πρόκειται να μας ε, δώσουν τη γνώμη τους ε, και αυτό θα βελτιώσει το κείμενο. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ δυναμικό το μήνυμα προς το Συμβουλίο. Και ότι αναβαθμίζεται η Ευρώπη χωρίς να φύγεται η εθνική κυριαρχία. Θα ήθελα απλώ να σα ενημερώσω ότι η ψηφοφορία της γνωμοδότησης θα γίνει στις 8 Μαΐου στην Επιτροπή μας Και κυρίως το πέρα τη δημόσια συνεδρίασης Αύριο θα συνεχίσουμε στις 9 με τη δημόσια κρόση για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Σας ευχαριστώ που λάβατε μέρος στην συνεδρίαση μας.